Ε, Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η νέα ενεργειακή αγορά και ο σχεδιασμός αυτής. Δημόσια ακρόαση. Βήμα-βήμα δημιουργούμε την Ενεργειακή Ένωση. Και σχεδιάζουμε εκ νέου την αγορά και ο σχεδιασμός ο νέος αυτός αγοράς είναι πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχάς διότι η αγορά μας σχεδιάστηκε εδώ και 40 χρόνια. Ούτως ώστε να εφοδιάζει την αγορά από μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας, πυρηνικές ε, μονάδες, με μηχανές, ε, με συγγνώμη, με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν ανοιχτά καύσιμα και τα τελευταία 20 χρόνια αλλάζουμε τους πόρους τους ενεργειακούς και τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρώτα απ' όλα θα μπορούσε εν μέρη να παραχθεί και με το φυσικό αέριο άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε την αγορά μας και θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ε, εσωτερική ενεργειακή αγορά σημαντικότατο αυτό όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση τον Ιούλιο Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη νέα ενεργειακή αγορά και το σχεδιασμό της, ούτως ώστε να δούμε ε, τη σχετική νομοθεσία για την ενεργειακή αγορά, κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Διότι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα για σήμερα. Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. πώς θα γίνεται η μεταφορά της ενέργειας, η πώληση. Δεν είναι εύκολο πρόβλημα να λυθεί. Θα εκπονούσε επί του θέματος έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούσε να συμβάλλει και το Κοινοβούλιο. Ο κ. Βέρνερ Λάγκερ είναι εισηγητής για την έκθεση πρωτοβουλίας και θέλει να προτείνει κάποιες λύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σκοπό τη ακροάσεω είναι να μπορεί κάθε μέλος να ακούσει και να, να συμμετέχει σε συζήτηση με εμπειρογνώμονε πριν την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση του κυρίου Λάγκεν και πριν ψηφίσει στις 20 Μαΐου, 24 Μαΐου με συγχωρείτε, 24 Μαου η Ήτρε. Η ακρόασή μα θα κρατήσει περίπου 2,5 ώρε και θα χωριστεί σε δύο τμήματα η ακρόαση. Η καθεμία θα καταλήγει σε ερωταπαντήσεις, περίπου 30 λεπτά. Οι εμπειρογνώμονες έχουν το πολύ 10 λεπτά χρόνο ομιλίας. Είναι ένα στενό περιθώριο για σας. Θέλει πειθαρχία αγαπητοί φιλοξενούμενοι και τα μέλη θα παρακαλούσα να περιοριστούν σε 2-3 λεπτά το πολύ. Θα δούμε πώς θα πάει. ούτως ώστε να αφήσουμε και χρόνο να δοθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν. Αν έχει την καλοσύνη να ξεκινήσετε τη συζήτηση, προβαίνοντας τα σχόλιά σας, εκφράζοντας τη γενική σας άποψη επί του ζητήματος. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, γερμανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για τη δημόσια κρόαση, καν για τη διεξαγωγή της. Είναι σημαντικό όταν εμεί νομοδοτούμε ε, και προετοιμάζουμε τις επόμενες νομοθεσίες να ακούμε τη φωνή των εμπειρογνωμόνων και των ειδικών. Όχι μόνο με γραπτές νομοδοτήσεις, αλλά να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και με τους ιδίους. Και θέλω να ευχαριστήσω ρητά το πρώτο πάνελ που δέχτηκε την ε, πρόσκλησή μας και ήρθαν για να συζητήσουμε. Η πρώτη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει παλιώσει λίγο, ήταν 15 Ιουλίου του 2015. Το Κοινοβούλιο ανέθεσε ε, την έκθεση στο δεύτερο ήμιση ε, του 2015 και το σχέδιο έκθεσής μου για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Στο μεταξύ είναι έτοιμο εδώ και λίγες εβδομάδες σε όλες τις γλώσσες. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, προσανατολισόμαστε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εξηγήσει που ήδη έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένα σημεία τονίζονται ε, για τους ε, εμπειρογνώμονες και εκείνους που ασχολούνται με το θέμα έχω να πω το εξής εισαγωγικά. Ξέρετε ότι στις πρώτη έκθεση, το σχέδιο έκθεσης έχουμε περιορισμό σε χαρακτήρες στην έκθεση. Δεν έχουμε βάλει όλα τα θέματα λοιπόν στο πρώτο σχέδιο. Θα ανοίξει ε, προθεσμία για τις τροπολογίες μετά την ακρόαση την άλλη εβδομάδα και μετά ε, τις διακοπές του Πάσχα των Καθολικών θα ακούσουμε και τους λεγόμενους ε, σκιώδεις ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων. Θα κάνουμε και την πρώτη μας λοιπόν ανταλλαγή απόψεων και μετά θα έρθει το θέμα στην Επιτροπή μας. Αυτά τα λέω εισαγωγικά. Ανασχεδιασμός λοιπόν της ε, αγοράς ενέργειας είναι ένας στόχος δεδηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί μία 20 έτη, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90 ακόμα ιδιαίτερα στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά μετά αργότερα και στο φυσικό αέριο. Είχαμε την αποδέσμευση, το unbundling. ο βασικός στόχος σήμερα του ανασχεδιασμού είναι ε, απότερος και το έχει ορίσει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού μας και ε, περιφερειακή συνεργασία θέλουμε να είναι πιο στενή στην ενεργειακή πολιτική, ιδιαίτερα σε επενδύσεις, σε νέες ε, καταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ε, διασυνδέσεις και ένταξη των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ενέργειας. Βέβαια αυτό το θέμα των ανανεώσιμων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτό, ακόμα και αν η αγορές σήμερα ενέργειας ε, διέπονται από εθνικά κριτήρια ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα που έχει κάθε χώρα και τους στόχους που έχει αυτή. Άρα λοιπόν η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι σωστή και το Κοινοβούλιο Ενδιαφέρεται πάρα πολύ, άλλωστε φάνηκε αυτό από τη μέχρι τώρα συζήτηση, να προωθήσει αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση όπως την έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πηγές παραγωγής ενέργειας. Δεν θα υπάρξει καμία σύσταση να καταργηθεί καμία μορφή παραγωγής ενέργειας, ούτε ο άνθρακας ούτε η πυρηνική ενέργεια ούτε πρόκειται μονομερώς να προωθηθούν ε, ε, κάποιες μορφές ενέργειας. Αλλά η προώθηση φυσικά των ανανεώσιμων είναι κάτι που κυριαρχεί και υπάρχει και το επίμαχο ζήτημα σε ποιο βαθμό οι εθνικοί μηχανισμοί ε, χωρητικότητας είναι απαραίτητοι ή τουλάχιστον προσωρινά ή μήπως θα μπορούσαν και να βλάψουν και να εμποδίζουν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η τάση των κρατών μελών έχει αυξηθεί να παίρνουν αποφάσεις σε 7 από 28 κράτη-μέλη ήδη ως προς το δυναμικό και τους μηχανισμούς χωρητικότητας, γιατί ε, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι στοιχείο που στο δινικές θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Η καλύτερη προϋπόθεση λοιπόν για καλύτερο ανεφοδιασμό είναι η συνεργασία ευρωπαϊκή, γι' αυτό ε, οι κρατικές παρεμβάσεις θα πρέπει να περιορίζονται κάθε είδους και να μην πω ότι πρέπει να ε, μειώνονται. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη η ενίσχυση πρόθεση ε, λόγω Τη απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων και θυμάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο άρχισε μια διαδικασία προσέφυγε κατά της Γαλλίας. Ξέρετε την πρόταση, ξέρετε τις διαδικασίες, το Κοινοβούλιο τα συζητάει όλα με ειλικρίνεια και τελικά εδώ στο όργανο αυτό που λέγεται Επιτροπή Βιομηχανίας θα πρέπει να έχουμε μια κάπως κοινή γραμμή για να κάνουμε συστάσεις στην Ολομέλεια. Και αυτό είναι ιδιαίτερη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρόπος λειτουργίας. Να σας πω λοιπόν τα βασικά της κεντρικής Ε, Οι διατιμημένες τιμές θα πρέπει και οι ρυθμιζόμενες να καταργηθούν. Τι γίνεται με τους διαχειριστές των δικτύων, πώς μπορούμε να συνδέσουμε την πρόθεση και ενίσχυση ε, τον ε, ΑΠΕ με τη σημερινή κατάσταση και να το διαχωρίσουμε από τις μόνιμες επιδοτήσεις. Ε, ποιος ο ρόλος που αναλογεί στους διανομής και τους διαχειριστές. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί πρέπει να εισάγουμε ένα καθεστώς ιδιοκτησίας όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παρόχους και τους διανομής. Θέλω να κλείσω εισαγωγικά. Βλέπω έχω ξεπεράσει κατά ένα το χρόνο μου, Πρόεδρε. Και σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σικητά. Τα πρώτα σας σχόλια θα ακολουθηθούν από συζήτηση. Πρώτος ομιλητής στο πάνελ. Ο πρώτος. Ξέρετε πολύ καλά ότι δημιουργούμε την εσωτερική αγορά αυτή για τους καταναλωτές μας, για τη βιομηχανία, για την οικονομία. Αλλά χωρίς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και πλατφόρμες εμπορίου ηλεκτρική ενέργειας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να δημιουργηθεί για αυτούς. Και στο τέλος τη διαδρομής η επιτυχία θα ανήκει, θα, θα οι πολίτες μας από αυτή. Πρώτος ομιλητής, ο Δόκτωρ Άλμπα Ρίος πρόεδρος της Euroelectric Market Committee Επιτροπή Επιτροπής Αγοράς. Euroelectric είναι το μεακό σύνδεσμος, ε, εκπροσωπεί τους φορείς της ηλεκτρικής Βιομηχανία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα του, στην Ισπανία, ο Δόκτωρ Αλμπαρίος είναι αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων της ΕΝΤΕΣΑ. για να παρουσιάσει το, τη θέση του ενεργειακού τομέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη δημιουργία της αγοράς και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ήτρε που μας προσεκάλεσε να συμμετάσχουμε σε αυτή την ακρόαση. Θα ξεκινήσω αναφερόμενο στο λογαριασμό του πελάτου. Αυτό είναι το α και το ω αυτόν που θα συζητήσουμε. Αυτό το γράφημα σας δείχνει πώς ο πελάτης, πώς ο λογαριασμός ενός ευρωπαϊκού νοικοκυριού έχει αλλάξει στην περίοδο 2008 μέχρι το 2014. Σε αυτό το λογαριασμό πληρώνουμε βασικά τρία πράγματα. Όλοι οι πελάτες πληρώνουν τρία πράγματα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού. Από τη μία πλευρά πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια αυτή καθεαυτή. Το κόστος παροχής ε, της ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουν και το δίκτυο για την διανομή και της ενέργειας που φέρνει την ενέργεια στα σπίτια τους. Και στο τρίτο πληρώνουν φόρο και το κόστος των πολιτικών. Διάφορα πράγματα είναι αυτά που πληρώνονται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού και που δεν σχετίζονται άμεσα στην, ε, στον εφοδιασμό, στην παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και βλέπουμε μεταξύ του 2008 και του 2014 το κόστος ε, εφοδιασμού στην ηλεκτρική ενέργεια μειώθηκε 5%, αυξήθηκε το κόστος του δικτύου κατά 18% και φόρος και, και πολιτική αυξήθηκαν κατά 47%. Και το κόστος εφοδιασμού σε ενέργεια μειώθηκε κατά 7%. Συγγνώμη. Κατά μέσο όρο πάνω από 1 τρίτο, δηλαδή 36% που πληρώνει ο πελάτης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού του, αποτελείται από φόρους και κόστος διαμορφώσεως πολιτικής σε κάποιες χώρες. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Στη χώρα μου, στην Ισπανία, είναι περίπου 50%. Στη Δανία είναι παρόμοιο ποσοστό. Στη Γερμανία πολύ ψηλό. Σε κάποιες χώρες, λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτή η φόρη και το κόστος της πολιτικής, αυτή η συνιστόσα που αυξάνεται μετάχιστο ρυθμό, σημαίνει ότι γίνεται ακριβώς ο ηλεκτρισμός με τεχνητό τρόπο και αυτό είναι ένα πρόβλημα διότι η ηλεκτροδότηση, ο εξηλεκτρισμός είναι ένας τρόπος να ε, βγάλουμε τον άνθρακα από την οικονομία. Αν θέλουμε να φύγει ο άνθρακας από την ενέργεια, από το ενεργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι τώρα, πρέπει να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα από την ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά, στη βιομηχανία και στις ε, μεταφορές και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν παράγει ε, εκπομπές άνθρακα. Αν γίνει ακριβή ηλεκτρική ενέργεια θα προτιμήσει ο πελάτης να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο για να θερμάνει την κατοικία του. Και αυτό δεν είναι λογικό από πλευρά ζησιμότητα, διότι θα χρησιμοποιούν οι πελάτε πετρέλαιο, ε, θα, αυτοκίνητα με διζελοκινητήρα αντί ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αυτό δεν έχει νόημα. Λοιπόν, αυτό το κόστος των φόρων και διαμορφώσεις πολιτικής ακριβένουν με τεχνητό τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια και κάνουν τους πελάτες να βλέπουν να αυξάνεται το πάγιο κόστος στο λογαριασμό τους που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και δεν μπορούν να αντιδράσουν σε αυτή την αλλαγή των τιμών της αγοράς. Λοιπόν, τώρα αν δούμε ποια είναι η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό της διαμάσης πολιτικής προσέρχεται από την υποστήριξη των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, διότι υποστηρίζουμε πολύ τις ε, ΑΠΕ. Ο στόχος της αναπτύξεως των ΑΠΕ είναι ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό έχουμε καθορίσει. Τελικά όμως τα περισσότερα, οι περισσότερε ΑΠΕ μπαίνουν στο σύστημα τη ηλεκτροδότηση και το μεγαλύτερο κόστο ανάπτυξη των ΑΠΕ πληρώνεται από του καταναλωτέ ηλεκτρική ενέργεια και όχι από αυτού που καταναλώνουν πετρέλαιο ή φυσικό φυσικό αέριο. Και έτσι ακριβένει η φυσικο αεριο ενέργεια. Λοιπόν, πρώτο μάθημα που μπορούμε να λύσουμε από εδώ. Αν γνωρίζουμε ότι αυτό το κόστος ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι πολύ υψηλό αν ξέρουμε ότι στο σύστημα το μελλοντικό με χαμηλό άνθρακα στο μέλλον θα έχουμε σημαντικό ποσοστό ΑΠΕ, σημαντικότερο από τώρα, καλύτερα να καταφέρουμε αυτές τις ΑΠΕ να τις κάνουμε αποδοτικές και ανταγωνιστικές. Τι σημαίνει αυτό κατά την απόψή μας. Ότι θα πρέπει οι ΑΠΕ να ενταχθούν στην αγορά, χρειάζεται ενίσχυση του συστήματος ανταλλαγής ρήπων, εμπορίου ρήπων, το ETS, ούτως ώστε να έχουμε ένα να στείλουμε ένα μήνυμα, να, να τονώσουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τα, οι μηχανισμοί που στηρίζουν τις ΑΠΕ και οι μελλοντικέ θα εδράζονται επί της αγοράς, θα είναι αποτελεσματικά συστήματα και θα εγγυώνται ότι θα οδηγούν σε μια ανταγωνιστική ε, εναλλακτική μορφή ενέργειας. Τι είδαμε λοιπόν στο προηγούμενο γράφημα, είδαμε το κόστος του δικτύου και αυξήθηκε το κόστος του δικτύου κατά 18% λαμβάνοντας υπόψη το πώς οι οικονομίες μας και οι κοινωνίες μας ε, εξελίχθηκαν και αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το, δίκτυο, το κόστος του δικτύου σχεδόν παρέμεινε σταθερό αν το λάβουμε αυτό υπόψη. Ε, και είναι λογικό αυτό, διότι η ρύθμιση των δικτύων μας εστιάζεται επί ελέγχου των επενδύσεων, επιμειώσεως του κόστους και μεγαλύτερης αποδοτικότητας και απλούστευσης. Πιθανότατα όμως δεν έχουμε τονίσει τα σωστά στοιχεία. Αν θέλουμε να εντάξουμε τις ΑΠΕ, αν θέλουμε οι πελάτες να αντιδρούν στα μηνύματα της αγοράς, αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ηλεκτροδότησης βιώσιμου, θα πρέπει να έχουμε δίκτυα τα οποία είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένα, πολύ πιο ευφυή από ό,τι είναι τώρα. Αυτό απαιτεί επενδύσεις, απαιτεί καινοτομία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί για τα δίκτυα ε, δεν δίνουν επαρκή κίνητρα για καινοτομία, επαρκή κίνητρα για αυτοματοποίηση του δικτύου, δεν δίνουν αρκετά κίνητρα για τη μεταμόρφωση που απαιτείται στο σύστημα ε, διανομής ε, και μετάδοσης, ούτω ώστε να ενταχθούν οι ΑΠΕ και τελικά το όλο σύστημα να είναι χαμηλό όσον αφορά τι και κατανάλωση άνθρακα. Μετά είναι για τον εφοδιασμό, για το, ε, επόμενο κομμάτι θυμής Βλέπετε η τιμή χοντρικής στη Γερμανία στην περίοδο 2009-2016. Μειώνεται, μειώνεται συνεχώς σχεδόν. Έχουμε επίπεδα τιμών τώρα που είναι ανάμεσα στα 20-25 ε, με 30 ευρώ ένα μεγαβάτ. Αυτό ε, δεν οδηγεί, δεν προσελκύει επενδύσεις, ε, δεν λαμβάνονται αποφάσεις περί επενδύσεων αποδοτικές, δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα για ανάπτυξη του συστήματος, δεν στέλνουμε μηνύματα για ανάπτυξη ιασδήποτε τεχνολογίας παραγωγής, ούτε θερμικής παραγωγής, ούτε με ΑΠΕ. Με αυτές τις τιμές δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα. Υπάρχει, υπερβολική, υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής. Αυτό είναι, ισχύει σε κάποιες χώρες. Έχουμε πολλή ενέργεια στο σύστημα, αλλά θέλουμε ακόμα να έχουμε δυνατότητα παραγωγής που να υπάρχει όταν δεν υπάρχει άνεμος, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια φερρυπίν. Και θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα, το δυναμικό και με αυτές τις τιμές που έχουμε σήμερα δεν θα δημιουργηθεί η δυνατότητα να έχουμε περιθώρια, περίσευμα ενέργεια στο δίκτυο. Ένα από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να υπάρξει δυναμικό ποσότητα να έχουμε την ενέργεια είναι ένα, ε, μια εύρυθμη ε, λειτουργία της αγοράς χοντρική και ένα από τα στοιχεία για να λειτουργεί αυτή η αγορά καλά είναι ε, οι τιμές όταν υπάρχει σπάνις, όταν υπάρχει έλλειψη εφοδιασμού θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές. Προφανώς αυτό είναι θεμελιώδες βασικό στοιχείο μιας αγοράς όταν υπάρχει έλλειψη προσφοράς να ανεβαίνουν οι τιμές. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Αυτές οι τιμές έλλειψης δεν υπάρχουν διότι υπάρχουν ανώτατα όρια που καθυστερούν τις αγορές και εμποδίζουν την αύξηση των τιμών της αγοράς να φτάσει στα επίπεδα που θα απαιτεί το. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε όμως σε ποιο βαθμό αυτές οι τιμές ε, έλλειψες ε, είναι οι σωστές και αν εξελίσσονται σωστά. Έχουμε ε, δύο ελλείψεις ασφαλείας εφοδιασμού έχουμε αυτές τις τιμές σπάνιδος ε, εφοδιασμού. Είναι πολιτικά αποδεκτό αυτό. Συμφωνούμε ότι περισσότεροι ότι πρέπει να έρθουν αυτά τα νότα τόρια των τιμών. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα, διότι τα νότα των τιμών πολύ, πολύ σπάνια τα φτάνουν οι τιμές. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το πρόβλημα. Παραγωγή που υποστηρίζεται, επιδοτείται, πολλή ενέργεια που δεν εξαρτάται από τιμές της αγοράς για να επιβιώσει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι τιμές έλλειψης δεν θα διαμορφωθούν. Η αγορά δεν θα φτάσει τα επίπεδα των τιμών έλλειψη ενέργειας. Άρα το επενδυτικό μήνυμα δεν αποστέλλεται και δεν δημιουργούνται οι αναγκαίες ευκαιρίες. Βασικά αυτές οι τιμές έλλειψης, ακόμα και αν είναι απαραίτητες, ακόμα και αν θέλουμε να αφαιρέσουμε τις τρευλώσεις που υπάρχουν, σπάνια αρκούν σαν κινητήρια δύναμη για επενδύσεις. Και σας προκαλώ να βρείτε επενδυτές, εταιρείε παραγωγής που είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε παραγωγή ε, βασιζόμενες στην έλλειψη ενέργειας αποκλειστικά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι εν γέννη η αγορά της ενέργειας πρέπει να συνδυάζει τρία στοιχεία. Χρειαζόμαστε μια αγορά για την ενέργεια, αυτή που έχουμε, αγορά για ευελιξία ούτω ώστε η δυνατότητα παραγωγής να μπορεί να προσαρμόζεται στι ανάγκες τη ζήτησης και τούμπαλιν και σε κάποιες περιπτώσεις όπου αυτό αρμόζει χρειαζόμαστε αγορά αποθήκευση δυναμικού να παράγεται η ποσότητα που χρειάζεται και να στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα για επενδύσει. Πρέπει να είναι ευρωπαϊκέ οι αγορέ, και Θα πρέπει να, είναι, ε, να σε ε, κοινέ αρχέ σχεδιασμού θα μπορεί να υπάρχει συμμετοχή σε διασυνοριακό επίπεδο κλπ. κλπ. Τώρα η περιφερειακή πτυχή είναι θεμελιώδης. Πιστεύουμε ότι φερειπίν οι τιμές έλλειψης και οι επάρκειες οι περιφερειακές είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποφασίσουμε κατά πόσο το σύστημα, συγκεκριμένη περιφέρεια, αν η αγορά δίδει αυτά που απαιτούνται και κατά πόσο χρειαζόμαστε και κάποιο άλλο στοιχείο, όπως μια αγορά αποθήκευσης ενέργειας και αυτό θα πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Η αξιολόγηση επαρκείας που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση της αγοράς που θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν το σύστημα, που είναι επιφορτισμένοι με αυτή την ανάλυση και που πρέπει πραγματικά να ασχοληθούν με την πραγματικότητα των επενδυτικών αναγκών. Επίσης, η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να συντονίζεται και να ολοκληρώνεται και σε περιφερειακό επίπεδο. Το τελευταίο σημείο που έχω να πω, όταν έχω μια αγορά δυναμικού εφοδιασμού, θα μου πείτε εκεί θα αυξηθούν οι τιμές. Δεν θα έπρεπε. Αυτή η αγορά, αν σχεδιαστεί σωστά, θα δίνει δυνα... τιμές δυνα... δυναμικού σε μηδέν αν υπάρχει μεγάλο δυναμικό και είναι μια ασφάλεια αυτή αν θέλετε και αντι... Ε, τελικά τις μεταβολές των τιμών έλλειψης τις μετατρέπει σε τιμές πιο σταθερές που μετατρέπονται σαν μήνυμα για επενδύσεις. Αν σχεδιαστεί σωστά αυτή η αγορά δυναμικού δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, δεν θα σημαίνει αύξηση του λογαριασμού που πληρώνουν τελικά οι πελάτες μας. Ευχαριστώ. Θα είναι τώρα εκπροσωπή μάλλον την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ανανεώσιμων Ενεργειών. Πρόκειται για την διευθύντριά της, καθηγήτρια κυρία Φουκέ. η οποία συμμετέχει και στην δικηγορική εταιρεία Better Bitner Health στο γραφείο Βρυξελών. Άρα, πρώτα πρόκειται για την Ένωση Εθνικών ε, Παρόχων Ανανεώσιμων Ενεργειών και έχετε το λόγο κύριε μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Μπούσεκ, ευχαριστώ και εσάς κύριε Λάγκεν και εσάς κύριε και κύριοι. Μεγάλη μου χαρά που μπορώ να παρουσιαστώ σήμερα ενώπιον σας για να μιλήσω για λογαριασμό της ΕΡΕΦ, δηλαδή της Ένωσης των οργανώσεων των ανεξάρτητων παρόχων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιθυμούμε και τώρα και τους επόμενους μήνες ε, να σας ενισχύσουμε στην προσπάθειά σας, στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ένωσης γενικά, για την ανανέωση της αγοράς ενέργειας και για την ε, επίτευξη των αλλαγών όπου αυτό απαιτείται. Πιθανώς Ε, να μην βλέπετε καλά στα μικρά γράμματα του πίνακα. Θα όμως πρόκειται για την κατάσταση στη Γερμανία και η πηγή είναι το Ινστιτούτο Οικολογικών Μελετών και περνά τις διάφορες φάσεις ανά τεχνολογία. Βλέπετε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, ε, πηγές ενέργειας μάλλον, συνδέονται με το γερμανικό σύστημα και σιγά σιγά και με το ευρωπαϊκό. Έχουμε και το σχέδιό μας που υπαγορεύεται ότι θα πρέπει να κάνουμε όπως είπε και ο κύριος ε, ε, Λάγκεν θα καταθέσουμε στοιχεία από το σχέδιό μας αυτό για τη συζήτησή σας και ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε στο έργο σας. Από τη δική μας σκοπιά η... ο σχεδιασμός για το 2009 έως 2028 είναι και πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς ένα σημαντικό θεμέλιο και παράδειγμα του μεγαλύτερου προγράμματος promotion παγκόσμια που ξεκινά από διάφορες αφιτηρίες με συνδυασμό πολλών χωρών και ιδίως χάρη στις προσπάθειες του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Ποια, ποιες είναι οι συνιστώσεις που πρέπει να εξετάσουμε για το νέο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα διαφοροποιηθούν. Ένα από τα πράγματα αυτά, αλλά θα αλλάξουν βεβαίω. Κάπου που δεν διαφοροποιούμεθα είναι ότι χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε μια καλή ισορροπία στην αγορά και ε, ένα καλό σύστημα intraday. Δεν χρειαζόμαστε capacity markets, αγορές ε, ε, δυναμικότητας. Χρειαζόμαστε να πούμε με διαθρωμένο τόπο, τρόπο και με τρόπο που θα γίνει κοινωνικά αποδεκτός από τις χώρες μέλη μας να καταργηθούν σταδιακά οι παλές πηγές ενέργειας, είτε είναι πυρηνικές είτε είναι άνθρακος. Χρειαζόμαστε μια διαρθρωμένη όθηση προς τα εμπρός. Και ο ΕΡΕΦ θεωρεί ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μόνες τους, αλλά το Κοινοβούλιο να δώσει μια γερή όθηση όπως τότε που κάναμε το επόμενο βήμα μετά από την κοινότητα Άνθρακος και Χάλιβος. Κάτι το οποίο θα προσφέρει μια διάρθρωση στις ε, χώρες μέλη. Όταν ήμουν νέα, ε, ήμουν αξιωματούχος στο Αμβούργο και αντιμετωπίσαμε τότε την ε, κρίση της ναυπηγικής βιομηχανίας που πήρε μετά και την Πολωνία και ολόκληρη την αυτή της Βαλτικής μπάλα όπως λέμε σε απλά ελληνικά. Το ζήτημα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να μειώσουμε τις πλεονασματικές, τα πλεονασματικά δυναμικά και να τα ξεχωρίσουμε από τα καινούργια. Και αυτό είναι δύσκολο θέμα και γι' αυτό ε, έχουμε ε, πρόβλημα και με τις τιμές αλλά και με τη διάθεση για επενδύσεις σε, νέες, σε νέα δυναμικά παραγωγής. Συχνά λένε ορισμένοι ότι τώρα πια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από μόνες τους. Δεν χρειάζεται πλέον ε, κατά προτεραιότητα δράση για τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματο από διάφορες πηγές, δηλαδή υπέρ των ανανεώσιμων. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος να το αγγίξουμε, διότι για μας η πολιτική δέσμευση της οδηγίας 2009-28 ήταν η προβλεψιμότητα και σε πολλές χώρες μέλη έχουμε δεσμευτικούς στόχους και είναι κρίμα που δεν, τους έχουμε πλέον, δεν θα τους έχουμε πλέον ως εθνικούς στόχους μετά το 2028, εκτός εάν το ανατρέψει αυτό το κοινοβούλιο. Το πακέτο σταθερότητας περιείχε ορισμένα στοιχεία. Καλό σχεδιασμό, προβλέψεις, στόχους. Το δεύτερο ήταν οι μηχανισμοί ε, πρημοδοτήσεων κλπ. Το τρίτο ήταν ε, η δράση προτεραιότητας και ήταν συνδυασμένο και με την οδηγία ενιαίας αγοράς και με την ε, οδηγία περί αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Και μπαίνουν τα στοιχεία αυτά και στη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτά δεν έγιναν επειδή μας αρέσανε απλώς, αλλά επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντελήφθησαν και ανέλησαν πολύ καθαρά ότι για να υπάρχει αξιόπιστη και ασφαλής αφετηρία για την συμμετοχή των ανανεώσιμων ε, στα δίκτυα θα πρέπει να υπάρχουν εγγύσεις για τους ε, παραγωγούς τέτοιας ενέργειας ότι θα μπορούν δηλαδή να ε, συνδέονται με τα δίκτυα και να παρέχουν την ενέργεια που παράγουν για να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις της αγοράς όπως αντιμετωπίσαμε σε ορισμένες χώρες με μονοπωλιακές δομές οι νεοεσελθόντες αντιμετώπισαν την αγορά με δυναμικά τα οποία είχαν υποτίθεται καταργηθεί και συχνά όμως εξακολουθούσαν να λειτουργούν μέσα σε ολιγοπολιακές ή μονοπωλιακές συνθήκες και ενώ τη Γερμανία που γνωρίζω το παράδειγμα δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων ενεργειών εάν δεν είχαμε δώσει ε, κατά προτεραιότητα θετικές δράσεις υπέρ των ανανεώσιμων ενεργειών. Υπήρξε λοιπόν αυτή η ιστορία επιτυχίας. Μιλούμε και για τη χώρα του εισηγητού μας τώρα. Το 2014 φτάσαμε από το 2,6 στο 25% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και, και άλλες χώρες όπως Ιδία Δανία που τα πάνε πολύ καλά. Άλλες όχι τόσο σε ορισμένα τμήματα όπως η Γερμανία δεν πηγαίνει πολύ καλά στις μεταφορές και στην βιομάζα. Όμως κάπου υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι για να ξεφύγουμε από την ε, κατά προτεραιότητα ε, δράση, κατά την προτεραιότητα ε, διασύνδεση, θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην προσπάθεια αφαίρεσης του άνθρακα από την ε, βιομηχανία ενέργειας. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα υπεσχημένα του Παρισιού. Γι' αυτό ο ΕΡΕΦ σας ζητεί να είστε πολύ προσεκτικοί στο επόμενο βήμα που θα κάνετε. Βέβαια, επιζητούμε συνέχιση των ε, εθνικών συστημάτων στήριξη των ανανεώσιμων ενεργειών, αλλά θέλουμε και πολύ μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Όπω θα έλεγε ένα ε, νομομαθή, τώρα εγώ εργάζομαι για την ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία, ε, για θέματα συμφωνιών με όμορε χώρε. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη επανάσταση σε, σε πολλέ περι, περιφέρειε τη Ευρώπη. Να μην το σταματήσουμε αυτό. Αντίθετα, να συνοδεύσουμε την προσπάθεια αυτή όσο γίνεται καλύτερα. Κάτι που είναι πράγματι δύσκολο είναι ότι έχουμε χώρες οι οποίες έχουν υποχωρήσει θεωρώντας ότι δεν έχουν ίσως την απαραίτητη οικονομική δύναμη λόγω πιέσεων επίσης από την Τρόικα να τροποποιήσουν τους μηχανισμούς στήριξης των ανανεώσιμων ενεργειών, αυτά για μας είναι θλιβερά νέα, διότι χάνουν ευκαιρίες οι χώρες αυτές. Χάνουν στην πορεία προς τον εξυγχρονισμό χάνουν βιώσιμες πηγές ενέργειας και χάνουν επίσης δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης με τρόπο ιδιαίτερα βιώσιμο. Και αν δεν τα ανανεώσουν όλα αυτά θα είναι μια χαμένη υπόθεση για πολλά χρόνια. Θα πρέπει να στεκόμαστε λοιπόν πολύ επικριτικά ε, απέναντι σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ισπανία που έχουν δει ε, αντιστροφή της πορείας αυτής και που ε, αυτή η αντιστροφή της πορείας είναι διαιτητήριο για οποιαδήποτε επένδυση. Ήθελα επίσης να σας δείξω να σας δείξω, έλεγα, τι γίνεται στην αγορά για τις ανανεώσιμες. Παρόλο που πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει ιδεώδης αγορά. Η αγορά υφίσταται στρεβλώσεις Υπάρχει υπερβολικό ε, παλαιό ε, δυναμικό παραγωγής σε χώρες όπως ε, το Ενωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο σύστημα στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος με πολλές εχμές και χρειάζεται να εξετάσουμε εκεί πολύ το στοιχείο της ευκαμψίας ή της ευελιξίας. Νομίζω ήδη μακρηγόρησα. Πάντως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τρόπο οικονομικό, δηλαδή οικονομικά αποτελεσματικό. Γνωρίζετε ότι οι τιμές για τις επενδύσεις για ανανεώσιμες ενέργειες, για παράδειγμα υπεράκτες κλπ, είναι υψηλές. Χρειάζεται να κάνουμε τη σχετική προσπάθεια. Είναι μια κοινή αναζήτηση και πρέπει να στύψουμε τα μυαλά μας, να καταλήξουμε σε λύσεις για να διατηρήσουμε τις βιώσιμες αυτές τις λύσεις. Με τα λόγια αυτά σας ευχαριστώ. Thank you, Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ακολουθεί ο τρίτος ομιλητής, Dr. Tobias Paulun από το European Energy Exchange AG, ε, που είναι μία από τις ε, ηγετικές πλατφόρμες ε, στην ε, Ευρώπη, ίσως και η μεγαλύτερη ε, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι επικεφαλής στη στρατηγική και επίσης εσείς δεν πουλάτε μόνο ρεύμα, αλλά και άδειες δικαιώματα αγοραπολισίας, εμπορίας, εκπομπών ρήπων. Έχετε το λόγο, Δ. Πάουλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευγένεια που είχατε να μας ε, καλέσετε και ευχαριστώ και τον κύριο Λάγκεν για την εκπόνηση της έκθεσης που είναι αρκετά ε, πλήρης και, καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο. Ε, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές ιδέες ε, σχετικά με τον όμιλό μας ε, που, ασχολείται με εμπόριο ηλεκτρική ενέργειας και φυσικού αερίου και κάνουμε και τις βασικές δημοπρασίες ε, για την παροχή δικαιωμάτων ε, εμπορίας εκπομπών ρήπων και κάποια άλλα εμπορεύματα. Ε, εμείς δεν είμαστε ιδιωτική εταιρεία μόνο, αλλά και δημόσια αρχή. Και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις από το καθεστώς αυτό, τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Μεταξύ άλλων αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχουμε διαφάνεια, συγκεκριμένε τιμέ σε όλου όσοι ενδιαφέρονται και δεν είναι μόνο φορεί τη αγορά αλλά και το γενικό κοινό ε, και να αυξήσουμε την ε, ρευστότητα και τον ανταγωνισμό στις αγορές. Ε, χειριζόμαστε και τη βραχυπρόθεσμη αγορά ε, ηλεκτρικής ενέργειας, η Apex Spot, ίσως τη γνωρίζετε, είναι αυτή η εταιρεία που δίνει μέσα αναφοράς, αλλά έχουμε και πιο μακροπρόθεσμα ε, με συμβόλαια για συγκεκριμένες μέρες, μήνες, εβδομάδες, έτη, μέχρι έξι ε, έτη στο μέλλον. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία για την αγορά αυτή, δεν είναι μόνο θέμα ανταλλαγή, είναι ουσιαστική αγορά που λειτουργεί από σήμερα. Οι ανταλλαγέ. το 2015 είχαμε πάνω από 3.000 τεραβατόρες με συνολικό όγκο πάνω από 100 δις ευρώ που διακινήθηκαν. Καταλαβαίνετε για ποια τάξη μεγέθους μιλούμε και πόσο σημαντικό ε, ε, είναι οι πλατφόρμες αυτές να εποπτεύονται σωστά. Ε, και μπορούμε να ε, καθοδηγούμε την παραγωγή και την κατανάλωση και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να δίνουμε κάποια μηνύματα για το πού πρέπει να πηγαίνουν οι επενδύσεις. Στην έκθεση λοιπόν του κυρίου Λάγκεν, καλύπτονται αυτά τα θέματα, έχει λάβει τη σωστή κατεύθυνση και τη σωστή προσέγγιση για το σχεδιασμό της μελλοντική αγοράς και είναι προσανατολισμένη στην αγορά, ελεύθερη από πολιτική καθοδήγηση και μιλά και για το βραχυπρόθεσμο, το πιο ευέλικτο σχήμα και το πιο μακροπρόθεσμο. Χαιρόμαστε που ζητάτε ε, ενισχυμένη ε, περιφερειακή συνεργασία και φυσικά επέκταση του δικτύου που είναι κλειδί εκ των όνων κάνουν για να υπάρξει ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά. Θέλουμε να τονίσουμε και εμείς ε, την υποστήριξη των ΑΠΕ ε, που θα πρέπει να βασίζεται στην αγορά πάντα και να είναι συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιες είναι οι απαιτήσει λοιπόν, τα προπετούμενα που θεωρούμε εμεί εκ των όνου κάνευ για τον ανασχεδιασμό της αγοράς εργασίας. Ακούστηκε ήδη και η τιμή σε περίπτωση έλλειψης ενέργειας. Αυτό είναι βασικό στοιχείο καθοδήγηση της αγοράς, ε, μια ελεύθερη αγορά που έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια. Το βλέπουν όλοι οι παραγωγοί 24 ώρες 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα και σε πραγματικό χρόνο ε, αγοράζει και πολύ κάποιος ε, ε, ρεύμα και χειρίζεται την παραγωγή και την κατανάλωση. Όταν έχουμε αυξημένη τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό δεν επηρεάζει το τιμολόγιο του ηλεκτρικού για τον τελικό καταναλωτή μακροπρόθεσμα. Δεν λειτουργεί έτσι. Ε, ε, ε, υπάρχει ένας προγραμματισμός σε βάθος πολλών ετών για να προστατεύονται τιμές. Όσο πιο εύκολο είναι να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές βράχη πρόθεσμα, τόσο προστατεύονται βράχη πρόθεσμα, μάλλον μάκρο και μέσο πρόθεσμα και τελικά προς του καταναλωτή. Ωστόσο, η EX ως μια πλατφόρμα ενέργειας εκτός ε, αυτής της αγοράς έχει αναπτύξει και κάποια εργαλεία που επιτρέπουν την ε, ε, μετατροπή των σκαμπανεβασμάτων βραχυπρόθεσμα των τιμών σε μια πιο μόνιμη σταθερότητα. Οι αγοροπολισίες ε, μπορεί να έχουν ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά έχουν πάντα υπόψη τους τη μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση για τα σύμβολα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι κανένας επενδυτής δεν θέλει να αγοράσει ένα νέο εργοστάσιο, ας πούμε, ε, πρέ, ε, υποχρεωμένος να ξέρει πόσο θα κάνει το ρεύμα, ποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Αυτό δεν γίνεται, αλλά... όταν ε, πολλούμε τέτοιες ασφάλειες, ε, το σκαμπανέβασμα, οι μετατροπές, οι διακοιμάνσεις των τιμών ε, μπορούν να μεταφραστούν σε κάποια μακροπρόθεσμη ασφάλεια σχεδιασμού και προγραμματισμού. Και μπορεί κανείς να προβάλλει τη σημερινή κατάσταση στο μέλλον με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή του μερίδιου των ανανεωσίμων. Άρα εμείς ε, θέλουμε να δεσμευτούν και οι πολιτικοί και οι ε, ρυθμιστικές αρχές να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες που τους δίνει η αγορά για ένα κίνητρο, για μεγαλύτερη ευελιξία, βράχη πρόθεσμα και μεγαλύτερες επενδύσεις και ασφάλεια μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, θα πρέπει να βασιζόμαστε και σε μηχανισμούς παραγωγής ισχύω ε, περισσότερο από αυτό που, που λειτουργεί σήμερα. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι καλή η ενίσχυση των ε, ε, ΑΠΕ. Θα πρέπει να μπουν στην αγορά, αλλά θα πρέπει να σέβονται και τα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Σας είπα, Cap Futures είναι ένα από τα στοιχεία που πουλούμε, αλλά υπάρχουν και ε, άλλα εργαλεία στην αγορά που παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες, σε μεμονωμένους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπορούν να φέρουν αυτές τις τεχνολογίες πιο κοντά στην αγορά. Από την άλλη έχουμε και τις, τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρειάζονται να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, όχι με την ίδια ευελιξία που θέλουν οι ανανεώσιμες. Ε, μόνο έτσι θα συναντηθούν πλήρως η προσφορά με τη ζήτηση. Κάτι άλλο που δεν ανέφερε αρκετά ή που δεν λέει αρκετά η έκθεση είναι η σημασία διασυνοριακών και μεγάλων αγορών και ρευστών ε, για να μπορεί κανείς να συμμετέχει σε μια δημοπρασία. Όσο πιο μικρή και κατερματισμένη είναι η αγορά, τόσο πιο δύσκολο είναι αυτό, όσο και δύνατο. Χρειάζεται μια ρευστότητα ε, και σε επίπεδο μεγαλύτερο από ό,τι ζήσαμε τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Οι μεγάλε ρευστέ αγορέ είναι αυτό που χρειαζόμαστε και όχι οι μικρές. Γι' αυτό χρειάζεται φυσικά επέκταση του δικτύου, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όταν αυτή καθυστερεί ε, πρέπει να βρούμε ε, προσωρινά μέτρα εναλλακτικά χωρίς να καταλήψουμε ε, το δρόμο αυτό της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει ασφάλεια εφοδιασμού. Αν το δούμε αυτό από ευρωπαϊκό επίπεδο, φυσικά καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να έχουμε πιο αποδοτικές λύσεις και πιο φθηνές με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, από ότι αν έπρεπε ο καθένας να το κάνει ξεχωριστά σε εθνικό επίπεδο, ορίζοντας την ασφάλειά του. Υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες για στενότερη συνεργασία των κρατών μελών, εμείς το καλωσορίζουμε, αλλά θα ζητούσαμε και περισσότερο περιφερειακό συντονισμό, έτσι ώστε να μην το παρακάνουμε και να ε, ε, ξεπεράσουμε κατά πολύ την ισχύ που χρειάζεται. Και ε, η αγορά είναι ήδη ευρωπαϊκή. σε διάφορους τομείς και θέλουμε και μηνύματα για την τιμολόγηση και σήμερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει έλλειψη ισχύω ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάντα, όχι σε εθνικό. Λοιπόν, αυτά ως προτάσεις, αν θέλετε να τις λάβετε υπόψη για να ε, υλοποιηθούν και αν υλοποιηθούν και αυτά τα μέτρα που ζητάει η έκθεση, δεν χρειάζονται νέες ρυθμίσεις για τις μακροπρόθεσμες ε, αγοραπολισίες. Λειτουργεί σήμερα η αγορά, ο αριθμός των φορέων ε, που συμμετέχουν είναι υψηλότερο από ποτέ. Είναι πάνω από 400 οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις δικές μας και μόνο αγορές. Και φυσικά είναι και όλοι και περισσότεροι γιατί δεν συμμετέχουν όλοι ε, στην ε, ανταλλαγή αυτή, στο ανταλλακτήριο αυτό, αλλά παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τις ειδήσει αυτές από την αγορά, τα μηνύματα που στέλνει η αγορά και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Mm. Τρεις ομιλίες είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ομιλητές μας για τα σχόλιά τους, για την παρουσίασή τους και τώρα θα έχουμε το κομμάτι με τις ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά έχετε πολλή δουλειά με τις απαντήσεις που θα έχουμε δώσει και τα σχόλιά μας. Ο εισηγητής μας ο κύριος Λάγκε, έχετε το λόγο. Ναι, να αρχίσω με μια ερώτηση προς τον καθένα. Κύριε ε, ε, Δόκτωρ Αλμπαρίος, είπατε ότι όταν οι φόροι και τα πολιτικά μέτρα μειώνονται, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και το καλύτερο μέτρο έτσι ώστε συνολικά να έχουμε ε, λογικές τελικές τιμές καταναλωτού. Ταυτόχρονα όμως ε, κάνατε μια απαρίθμηση και μας δείξατε ότι Κατά τη δική σας άποψη το καλύτερο θα ήταν ε, να μην κοιτάμε μόνο το energy only, ε, μόνο ενέργεια, αλλά να έχουμε και κάποιες άλλες αγορές ε, ηλεκτροπαραγωγικών ικανοτήτων, ισχύως Capacity market δηλαδή αυτό λέγεται. Μα αυτό δεν είναι κάπως αντιφατικό. Θέλουμε από τη μια να βάλουμε τις ανανεώσιμες και από την άλλη να έχουμε εγκαταστημένη ισχύ για συγκεκριμένα παραδοσιακά συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Είπατε αυτό που έχει σημασία είναι η αποθήκευση. Ε, μα η αποζημίωση δεν έχει, ε, κυρία Φουκέ, Σημασία, μόνο η προτεραιότητα είναι αυτή. Και να ρωτήσω κάτι για το ανταλλακτήριο, το χρηματιστήριο τη ενέργεια, το Dr. Paul. Intraday εμπόριο λέγεται αυτό, μέσα σε μία μέρα. Ε, Μιλήσατε για τα μακροπρόθεσμα, τα μεγάλα στοιχεία και τα λοιπά, ωραία είναι αυτά, ε, τις μεγάλες συμβάσεις και τα μακρινά συμβόλαια. Τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο όμως, μέσα σε μία μέρα. Πώς, είναι η ψαλίδα ανάμεσα ε, στην ανάγκη και το εμπόριο, δηλαδή τη διάθεση. Το δικό σας χρηματιστήριο αυτό πώς το έχει δει. Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Κομπουλανέτσι. Thank you. Uh, thank you for the... Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ο κ. Αντωνάτος και όδης για το θέμα αυτό δεν είναι εδώ, οπότε δεν μπορώ να αναλάβω στη θέση του. Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα στην ομάδα είναι καλή βάση αυτή για την έκθεση τα καυτά θέματα. Η αγορά δυνατοτήτων του δυναμικού. Είδα. Οι ενεργειακές εταιρείε παραγωγής ενέργειας ήταν πρώτα να μην φορολογηθούν και μετά θέλουν να πάρουν εγγυημένα χρήματα. Βλέπω την αλλαγή παρετούμεθα από την, ελέξη την, αγορά, την οικονομία της αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια ή όχι. Έχουμε τα νότατα όρια κλπ. Και προσπαθούμε να δούμε τις διασυνδέσεις, το σχεδιασμό κλπ. για να θέσουμε τις ΑΠΕ να συμπεριληφθούν και να αντικαταστήσουν άλλες ενέργειες. Μόνο μηχανισμό μηχανισμός δυνατοτήτων θα δημιουργεί αυτό. Πιθανότατα θα υπάρξουν κάποια μοντέλα και κάποιες τεχνολογίες για να αποφευχθεί. Η δεμή θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είναι ανοιχτή η αγορά για φορείς διαφόρων μεγεθών, χρήστες διαφορετικών καυσίμων, θέλουμε αποδοτικότητα στην ενέργεια και να χρησιμοποιήσουμε τις ΑΠΕ. Εξ αρχής να πω ότι αυτό το θέμα, ο νέος σχεδιασμός αγοράς ενέργειας θα πρέπει να μετονομαστεί και να ονομαστεί νέο σχεδιασμό αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι αλήθεια, δεν μιλάμε για την ενέργεια και τι ενεργειακέ αγορέ. Εδώ ακούσαμε το γερμανικό παράδειγμα. Αν δείτε τη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια στο γερμανικό μοντέλο, χρησιμοποιείται η βιομάζα, ηλεκτρισμός. Uh, really the question there, do we want Europe to have the Θέλουμε να έχει... Τι, πώς θα αντιμετωπίσουμε ισορροπία σε όλη την Ευρώπη. Όποτε κάποιο τροφοδοτεί με ενέργεια το δίκτυο θα πληρώνεται ακόμα και αν δεν χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το σύστημα. Είμαστε, έρχομαι από την περιοχή που είναι στον αρκτικό κύκλο. Ε, υπάρχουν επιδοτήσεις, αγορά κλπ. Πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, τι ανάγκες υπάρχουν για κάθε περιοχή. Τελικά σχόλια. Το ιδεώδες θα ήταν να απαλλαχθούμε από όλες τις επιδοτήσεις. Ακόμα υπάρχει κάποια ανάγκη για αυτές. Ίσως δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Ίσως χρειαζόμαστε φυείς επιδοτήσεις. Βάση περιφερειακών αναγκών. Να χρησιμοποιούμε το νερό όποτε χρειάζεται, βιομάζα όποτε χρειάζεται κλπ. Ίσως να αλλάξουμε τον τίτλο. Uh, uh, uh, ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ, λέει ο Στυλίτσκα, για τις παρουσιάσεις σας. Καταρχάς, εκτιμώ το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Λάγκε, στηρίζεται στους σωστούς πυλώνες. Εξετάζουμε την αγορά ενέργειας ή της ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες. Αν ήμουν ιδιοκτήτης επιχειρήσεως. Δεν θα είχα κίνητρα κανέναν λόγο να επενδύσω. Αν κάναμε ένα γράφημα, γραφική παράσταση, δεν θα βρίσκαμε κάποιον τομέα όπου θα ήταν οικονομικά βιώσιμο να επενδύσει κανείς όσον αφορά την ενέργεια. Δύσκολο να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Ήγηκε η ώρα και έπρεπε να γίνει πιο πριν. Μέσω τη εκθέσεως να δώσουμε όθηση σε εμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενό σχεδιασμού. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειε. Θα έχω κάποια σχόλια στον αφορά το σχέδιο εκθέσεως. Για την ώρα θα πω ότι οι βασικές αρχές με βρίσκουν σύμφωνο. Ίσως πρέπει κάπου να συμπληρώσουμε κάποια σημεία, να ενισχύσουμε κάποια σημεία. Εν γέννη όμως Συμφωνώ. Εκμεταλλεύομαι την παρουσία σας θέτοντας ερωτήσεις. Από τον κύριο Αμπάριος. Δεν αναφερθήκατε στις διάφορες ζώνες εσείς. Ζώνες δημοπρασίας. Προβλέπω τι θα πείτε, αλλά αν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σας παρακαλώ. Κύριε Μπαρίας, αναφερθήκατε στο μηχανισμό δημιουργίας δυναμικού παραγωγής. Κατάλαβα τη θέση σας. Ποιο λεπτομερή απάντηση μπορείτε να μου δώσετε. Θέση πιο λεπτομερή. Είναι έσχατη, με το έσχατη ανάγκης. Ποια είναι τα κριτήρια. Υπό οποίες προϋποθέσεις. Και για πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν αυτές οι αγορές δυνατοτήτων. Και στο συνάδελφό σας θέλω το ίδιο ερώτημα. Οι επιδοτήσεις αναφέρθηκαν. Καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι εννοείται προς τα που κινείστε. Είναι πραγματικότητα σήμερα. Συμβάλλουν στη στρέβλωση της αγοράς. Οι επιδοτήσεις αυτές καθ' αυτές και η κατάχρηση αυτών ίσως. Εγώ είμαι Τσέχος και μιλώ ανοιχτά. Με την ηλιακή ενέργεια διαπράξαμε απάτες. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα όμως για τις επιδοτήσεις σχετικά με αυτό. Έχω σαφέστατη στεναρή θέση από αυτού, αλλά θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Κυρία Φουκέ, αν κατάλαβα καλά, ποια είναι η θέση σας για την ένταξη των ανανεωσίμων στο σύστημα. Μπορείτε να μου δώσετε λεπτομέρειες. θέλατε να προωθηθούν οι ανανεώσιμες. Έχουν πλήρη υποστήριξη. Την πλήρη υποστήριξή μου η ΑΠΕ. Θα ήθελα όσον αφορά την ένταξή του στο δίκτυο του σύστημα να δω ποιον θέσαι. Ο κύριος Μαραγάλ έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Sí, Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πάνελ και αυτά που μας λέτε και ε, έτσι είχε και μεγάλη ποικιλομορφία γιατί ο καθένας εκπροσωπεί με μεγάλη πίστη και αφοσίωση τον κλάδο του ή το φορέα του και ε, αυτά που θέλει να υπερασπιστεί και να προωθήσει ε, και τα επιχειρήματά του. Πάρα πολύ σύντομα σε σχέση με τόσα υπόθηκαν. Οι μηχανισμοί παραγωγής ισχύω ε, είναι στρέβλωση για τις αγορές. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είναι η τελευταία καταφυγή και το τελευταίο σύνορο ενός συστήματος που ελπίζω να είναι σε αποδρομή και σε εξαφάνιση για την ασφάλεια ανεφοδιασμού, αλλά ουσιαστικά τι κάνει είναι κρυφές ε, ε, κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων αν είχαμε ένα καλό σχεδιασμό των περιφερειακών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύτερα από τα εθνικά, αυτό δεν θα χρειαζόταν. Και θα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ήδη υπερπαραγωγή και υπερβολική ισχύ. Υπάρχουν μηχανισμοί διασύνθεσης, υπάρχουν αρχές της ρευστότητα και της ευελιξίας, όλα αυτά καλά, αλλά υπάρχει υπερπαραγωγή τελικά στην ενέργεια ε, προς την ισχύ. Και θα το καταλαβαίναμε απολύτω αν είχαμε αυτή την περιφερειακή προσέγγιση. Για την ευελιξία. Μιλούμε για μια αγορά η οποία πρέπει να δώσει χώρο στις ανανεώσιμες. Εάν το κάνει αυτό θα σημάνει ότι οι πληστηριασμοί θα γίνονται και οι δημοπρασίες ε, όσο γίνεται πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο. Ε, τώρα ε, το έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά και με τις ανανεώσιμες θα μπορούσε να γίνει την ίδια μέρα και σε 15 λεπτά μέσα, σε ένα τέταρτο για να αγοράσει κανείς το ρεύμα που χρειάζεται, το επιπλέον. Εκατέρωθεν. Και όταν μιλάμε για την πλευρά της ζήτησης και τη διαχείριση από εκεί, είναι ο καλύτερος τρόπος, ίσως και ο μοναδικός, έτσι ώστε οι καταναλωτές, οι μεγάλοι, έτσι οι βιομηχανικοί ε, καταναλωτές, αλλά και τα μικρά νοικοκυριά, γιατί όχι, να ξέρουν πώς θα διαχειρίζονται το δίκτυό τους και ε, σε σχέση με τις μεταβολές και τις διασκημάσεις των τιμών. Για να ξέρει ο καθένας να κανονίζει την πορεία του, να παράγει, να καταναλώνει κτλ. Το ίδιο και όταν μιλάμε για δυναμική τιμολόγηση. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πρέπει οι τιμές να αντανακλούν την κατάσταση αν έχουμε έλλειψη ή πλεόνασμα ενέργειας. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν τα κατάλληλα μηνύματα προς τους ε, επενδυτές που μπορεί να είναι οι διεκτήτες του δικτύου ή πάροχοι ε, διανομής. Και ένα άλλο που θέλω να πω το εξή. Θα πρέπει να προσαρμοστεί και ο χάρτης, ο θεσμικός, να ενισχυθεί ο ρόλος του Acer, του ρυθμιστή, για να μπορεί καλύτερα να συντονίζει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ηλεκτρικής ενέργειας και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί φορείς θα πρέπει να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις εθνικές αρχές. Έχω να πω κι άλλα για ευρωπαϊκές επενδύσεις και δίκτυα κτλ. Δεν διέλειωσα. Ένα, ένα σχόλιο μόνο. Για την Εντέσα, την Ισπανική ΔΕΗ. Δέκα δεύτερα δεν μου δίνετε πρόεδρε. Εντάξει, δεύτερα, δέκα μόνο. Έλεγα λοιπόν, σε χώρες όπως η Ισπανία που είναι η πατρίδα μου, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στο διαχωρισμό του παραγωγού ε, και του ε, εμπόρου, του διακινητού του δικτύου, αλλιώς ε, στρεβλώνουμε, στρεβλώνουμε την αγορά. Το λόγο έχει η κυρία Ένστ, εξονομέτως της Γκουε. Um- Ευχαριστώ. Αυτό που μας βασανίζει εμάς το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο και μας ταλαιπωρεί. Πώς μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε έναν τύπο αγοράς που να είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετείται όλο και περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί βασίζεται σε αυτό. Πώς μπορούμε να ανασχεδιάσουμε έτσι την αγορά μας για να το πετύχουμε και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε οι αποφάσεις του Παρισιού για το κλίμα να υλοποιηθούν. Όλα αυτά είναι τα αποφασιστικά, αυτό μας ταλανίζει εμάς και θα πρέπει αυτό να είναι ε, και οικονομικά συμφέρον και να μπορούν να το επομίζονται και οι τελικοί καταναλωτές, να το πληρώνουν δηλαδή. Και ε, τρία πράγματα μας ενδιαφέρουν εδώ. Πρώτον, ο μηχανισμός παραγωγής ισχύω ή η αγορά, αυτό το capacity market, τι είναι ακριβώς, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ο πρώτος με τον τρίτο ομιλητή δεν συμφωνούν πάντα. Ε, ο μηχανισμός λοιπόν παραγωγής ε, δυναμικότητας ισχύω τι είναι. Και το λένε πολλά ερευνητικά Ινστιτούτα που το έχουν ψάξει λέει ότι εδώ μπορούν να υπάρχουν ε, προβλήματα στη ρυθμιστική αρχή ή δυσκολεύουν ε, το μετασχηματισμό των ενεργειακών ηλεκτρικών συστημάτων. Είναι δύσκολο να ενταχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν υπάρχει ένας μηχανισμός παραγωγής ισχύω. Υπάρχουν πολλές επικρίσεις και θα ήθελα να μου απαντήσετε. Να μου απαντήσετε παρακαλώ πώς το βλέπετε πολύ συγκεκριμένα. Χρειάζεται ακόμα κάποιος μηχανισμός παραγωγής ισχύω που να θεσπίζουν τα κράτη. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα ε, ασφάλειας εφοδιασμού ή θα πρέπει να ξεφύγουμε από οποιασδήποτε επιδοτούμενες παραγωγές ισχύω, όπως είπε η κυρία Φουκέ, να, να τα καταλήψουμε αυτά ή να τα καταστήσουμε από κάτι άλλο. Γιατί εμείς θα πρέπει να διαμορφώσουμε θέση και στάση. Δεύτερο, ε, εθνικά ενεργειακά μείγματα. Όταν λέτε από τη μια ότι δεν εξαιρούμε καμιά μορφή ενέργειας, πώς είναι δυνατόν να προωθούμε τις ανανεώσιμες. Θα παρακαλούσα την κυρία Φουκέ να μας απαντήσει πώς το βλέπετε. Και ένα τελευταίο τρίτο πολύ γρήγορα, οι επιδοτήσεις στις κρατικές ενισχύσεις. Είπατε κυρία Φουκέ μάλιστα, υπάρχουν τέτοιες και για τις ανανεώσιμες, υπάρχουν κάποια κίνητρα ή ε, εθνικά συστήματα ενισχύσεων και προωθήσεων. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Πάμε σε άλλου ομιλητέ. Όχι πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ. Η κυρία Ντεγκαστήγιο έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Λοιπόν, ναι, ισπανικά θα μιλήσω, βάλτε τα. ακούσαμε ε, κάτι που είναι προφανές. Εδώ έχουμε διαφορές από χώρα σε χώρα. Αυτό δεν, ακούστηκε, αλλά το αφήσατε να εννοηθεί. Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Κάθε χώρα σχεδιάζει την αγορά ενέργειας δικιά της. Και τώρα που βρισκόμαστε. Υπάρχουν καταστάσεις πολύ διαφορετικές που επικρατούν από χώρα σε χώρα, έτσι δεν είναι. Ορισμένοι έχουν αποκλειστικά σχεδόν πυρηνική ενέργεια, άλλες χώρες έχουν ένα μείγμα με πυρηνική ενέργεια, άλλες χώρες έχουν λάβει την απόφαση ότι όχι, φεύγουμε από τα πυρηνικά και μάλιστα στο προσεχές μέλλον δεν εγκαταλείπουμε τελείως την πυρηνική ενέργεια και το μείγμα προσανατολίζεται πολύ περισσότερο στις ανανεώσιμες πάνω από το μεσόρο τον ευρωπαϊκό. Υπάρχουν άλλες χώρες που δεν έχουν προβλήματα διασύνδεσης, ενώ κάποιες χώρες έχουν, οπότε δεν μπορούν να πούν ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας έλλειψης ε, ε, παροχής από τις διασύνδεσεις. Δηλαδή είναι τεράστιο ψηφιδωτό αυτό διαφορετικών καταστάσεων. Ο στόχος λοιπόν του σχεδιασμού ή του ανασχεδιασμού που θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν όλοι. Οι οι makers, εκείνοι που παίρνουν τι πολιτικέ αποφάσει, εκείνοι που είναι ενεχόμενοι και ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουμε ένα στοιχειώδη κοινό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να έχουμε ενιαίο και ομοιόμορφο. Λοιπόν, σε ένα στοιχειώδη ελάχιστο κοινό σχεδιασμό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κοινού στόχου, βεβαίω, απολύτω. Όπω είναι η εγκατάλειψη του άνθρακα, να ξεφύγουμε, να αποκυστρωθούμε από τον άνθρακα, η, η αύξηση σημασία και του μεριδίου των ανανεωσίμων πηγών ενέργεια, η ασφάλεια του ανεφοδιασμού ή του εφοδιασμού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Τελική τιμή καταναλωτού, γιατί τελικά ο καταναλωτής πληρώνει τα σπασμένα όλων των αποφάσεων που μας έρχεται εμάς να πάρουμε. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια στοιχειώδη ε, απόφαση για ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή σχεδιασμού που να είναι πρόοδος φυσικά σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και το ψηφιδατό. Κύριος κύριο <clears throat> Thank Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και τις και τους ομιλητές. Έχω ορισμένε ερωτήσεις, αλλά πρώτα ένα γενικό σχόλιο. Αφού συμφωνήσω με τον κύριο Αλβαρίος που είπε ότι όλα αρχίζουν από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί πρέπει να ε, στοχεύσουμε ιδιαίτερα. Με τον Βέρνερ πήγαμε και είδαμε τον διαχειριστή δικτύου άπριον και μας έδειξαν σε πίνακες τις πραγματικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι υπάροχοι ενέργειας, με τις ανανεώσιμες ενέργειες δηλαδή, όταν σταματούν να γυρνούν οι τουρμπίνες, οι ανεμογεννήτριες, διότι δεν φυσάει πια. Και μας έδειξαν στο δίκτυο πρόσφατο σταθμό παραγωγής θερμοηλεκτρικό που τελικά είχε απόδοση μηδέν διότι ήταν λιγό, πιο οικονομικό να μην λειτουργεί παρά να λειτουργεί. Κόστισε περισσότερο η λειτουργία του. Ε, λοιπόν πρέπει, η φυσική είναι φυσική και δεν αλλάζουν οι κανόνες της και οι τιμές δεν ακολουθούν, χρειάζονται επενδύσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την κυρία Φουκέ προς την και εν πάση περιπτώσει. Νομίζετε ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες και ότι αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός. Πώς ε, τότε θα ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των τιμών. Ε, Πήγα και είδα τον διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί την παραγωγή, το δυναμικό, όταν το ένα σταματάει και λειτουργεί το άλλο. Βλέπετε και αυτό είναι ο πραγματικό κόσμο. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε τώρα για του άλλου δύο μιλητέ, Ρίο και Πούλιν. Ποια είναι η διαφορά. Εσεί μιλήσατε πρώτα για capacity markets, ενώ ο τρίτο μίλησε για ένα είδο futures trading. Εγώ νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οι capacity markets είναι μετά από τρία χρόνια. Ποιε θα είναι οι τιμέ. Ε, ποια είναι η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στα δύο αυτά. Πάολ Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι μια από τις πραγματικές ερωτήσεις πρέπει να είναι εάν πραγματικά χρειαζόμαστε capacity markets θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνει αυτό μέσα σε μια πανευρωπαϊκή πρόσκληση εκδηλώσεως ε, ενδιαφέροντος για να δούμε και ποιος είναι αυτός ο, ο οποίος θα κάνει και τις καλύτερες προσφορές και για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις ε, ε, αγορές δυναμικού capacity markets. Δηλαδή εφόσον μεσοπρόθεσμα μπορούμε να, θέλουμε μάλλον να φτιάξουμε ε, μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, δεν μπορεί να υπάρχουν πλέον ζώνε εθνικών τυπών. Χρειαζόμαστε περιφερειακέ ζώνε οι οποίε τουλάχιστον θα υπερβαίνουν ένα τουλάχιστον εθνικό σύνορο. Διότι αν εφαρμόσουμε το παλαιό σύστημα, τότε στον τομέα αυτό δεν θα επιτευχθούν τίποτε σημαντικά βήματα πρόοδου. Η ερώτησή μου τώρα έχει ω εξή είπε και ο κύριος Κάρινς κάτι σχετικό, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ε, φυσικές αγορές, τις πραγματικές αγορές δηλαδή, με τις τιμές στα χρηματιστήρια. Πώς θα συμβαδίσουν τα πράγματα αυτά. Και τέλος, νομίζετε ότι για την εξέλιξη των εφιών δικτύων είναι αναγκαίο να συγχωνεθούν Άσα και Μπέρετς ή Μπέρεκ. για να μπορούν να γίνονται ε, οι σωστές διακινήσεις του ρεύματος. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Μπούσεκ. Θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε. ο Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Η αγορά ε, παραγωγής δυναμικού, παραγωγής ισχύω είναι κάτι απαραίτητο. Αυτή ήταν μια από τις ερωτήσεις των βουλευτών. Δεν υπάρχει μια και μοναδική απάντηση σε αυτό. Η κυρία Πιλάρντε Καστίγιο το εξέφρασε άριστα. Εξαρτάται. Εξαρτάται από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, από την κατάσταση της αγοράς, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Η αγορά ισχύω δεν είναι κάτι καλό ούτε κακό. Πρέπει να προβούμε σε ανάλυση κατά περίπτωση. Αυτή η ανάλυση είναι η ανάλυση επάρκειας όπως αποκαλείται. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις περιστάσεις που επικρατούν σε μια αγορά, περιφερειακή αγορά, όχι εθνική. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση της αγοράς, μια ανάλυση των τιμών, των δυνατοτήτων παραγωγής ισχύω, προσδοκίας παραγωγής, πώς μπορούν να επιβιώσουν οι δυνατότητες παραγωγής στις συνθήκες της αγοράς, πώς, ποιες προσδοκίες υπάρχουν για εξέλιξη της αγοράς και το καθεξής. Και το αποτέλεσμα της αναλύσεως θα αφορά το επίπεδο επαρκείας μιας συγκεκριμένης αγοράς. Τώρα τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν στόχους επαρκείας. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να πούν πόσο αξιοπιστία θέλουν να έχει το σύστημά τους. Και σχεδόν κανείς δεν τους, αρνείται το δικαίωμα. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν διαφανώς να το καθαρίσουν αυτό, να μπορούμε να, να συγκρίνουμε τα στοιχεία τα ίδια α, τις ίδιες μεταβλητές για να μπορούμε να συγκρίνουμε τους διάφορους στόχους των διαφόρων κυβερνήσεων και μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση σε μια δοθήσα αγορά αποτέλεσμα τέτοιας αναλύσεως σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι ότι χρειάζεται μια αγορά ισχύω. Όταν δημιουργηθεί έτσι μια αγορά, τι είναι, επιδότηση, είναι μια αγορά για διαφορετικό προϊόν που θεωρείται ισχύς, δυναμικό, είτε ενέργεια, ενέργεια και ευελιξία. Και χρειαζόμαστε στο σύστημά μας ισχύ. Αν θέλουμε να έχουμε μεγάλο ποσοστό ανανεωσίμων, χρειαζόμαστε μια σταθερή, σταθερό δυναμικό που πολλοί, πολλοί πάροχοι να δημιουργούν αυτή την παραγωγή ισχύω. Γι' αυτό πρέπει η αγορά ισχύω να μην είναι μόνο ανοιχτή σε αυτού που παράγουν την ενέργεια, σε αυτού που αποθηκεύουν, αυτού που χειρίζονται την ενέργεια, διότι όλοι αυτοί οι φορεί μπορούν να δώσουν σταθερότητα και να αντιδράσουν στι ανάγκε ισχύω ε, του συστήματο. Αυτό δεν είναι επιδότηση, είναι ένα άλλου είδου αγορά δημιουργείται σε διαφορετική χρονική στιγμή αυτή η αγορά ε, για διαφορετικούς σκοπούς. Τώρα το προϊόν αυτό είναι κάτι τρελό. Ας σκεφτούμε στο μέλλον. Πάμε στο 2050. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τον άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το σύστημα του μέλλοντος λοιπόν πιθανότατα σε πολλές χώρες θα είναι 100% Ανανεώσιμε σύναποθήκευση. Σε κάποιε χώρε θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια άλλη τεχνολογία ή πυρηνική. Πιθανότατα σε πολλέ χώρε θα έχουμε ένα σύστημα με ανανεώσιμε συν αποθήκευση. Βασικά θα αποτελείται από παραγωγή με σημαντικό κόστος επενδυτικό και βασικά καθόλου μεταβλητό κόστος. Ένα σύστημα όπου η πυρηνικη πιθανοτατα σε πολλε χωρε θα εχουμε ενα συστημα με ανανεωσιμε συν βασικα θα αποτελειται απο παραγωγη με σημαντικο κοστος επενδυτικο και βασικα καθολου μεταβλητο κοστος ενα συστημα οπου η τιμη του καυσίμου δεν είναι σχετική, διότι χρησιμοποιούμε καύσιμο και διοξιδίου του άνθρακος η τιμή δεν έχει σχέση, δεν παράγουμε διοξιδίου του άνθρακος. Το σύστημα αυτό, η δομή του κόστους είναι πάγιο κόστος βασικά. Αυτό ακριβώς έχουμε τώρα στις τηλεπικοινωνίες. Εδώ και κάποια χρόνια πληρώναμε τηλεπικοινωνίες βάσει των διαβιβαζομένων πληροφοριών ή βάση του χρόνου χρήσεως. Τώρα κανείς δεν κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ έχω ε, εύρος συχνοτήτων συγκεκριμένων στη χώρα μου και κανείς δεν μου λέει πόσες πληροφορίες θα φέρω στο σπίτι μου αν οι πληροφορίες χωρούν στο εύρος της ζώνης. Στο μέλλον θα είναι παρόμοιο και το σύστημα ενεργείας και η μεταβλητή θα είναι ισχύς. Θα πρέπει να έχουμε μια αγορά που σχεδιάζεται και μας κατευθύνει προς αυτή την αντιμετώπιση. Ετέθη ε, ε, ένα ερώτημα όσον αφορά τιμολόγηση. Αυτό προβληματίζει κυρίως τη τσεχική δημοκρατία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Θα πρέπει ότι θέλουμε ρευστότητα και ε, ανταγωνισμό. Το μέγεθος των ε, πληστηριασμών χρειάζεται τη σωστή ε, δομή της διάφορες ζώνες. Εξαρτάται από το κόστος και τη δομή του δικτύου και δεν μπορούμε να έχουμε ε, ζώνη δημοπρασιών που περιορίζεται πολιτικά αλλά από φυσικά και τεχνικά ε, όρια. Υπάρχουν διαδικασίες που θεσπίζονται στον κώδικα των δικτύων που καθορίζει το μέγεθος της ζώνης χρεώσης και πώς αυτές θα πρέπει να αλλάζουν όταν εντοπίζεται ότι δεν λειτουργούν σωστά. Υπήρξε ένα ερώτημα για την αγορά ισχύω έναντι των futures. Υπάρχει αγορά futures αυτών των αξιογράφων που μπορώ να πουλήσω ενέργεια ε, δύο-τρία χρόνια πριν. Όχι με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Αν γίνει οι περισσότεροι επενδυτέ, θα έλεγα όλοι οι επενδυτέ, θα θεωρήσουν ότι αυτό δεν αρκεί για επενδύσει. Αυτοί οι επενδυτέ χρησιμοποιούν ε, ε, ένα πιο μακρινό ορίζοντα χρονικά και δεν μπορούμε να επενδύσουμε γνωρίζοντα το κόστο του επομένου χρόνου ή το κόστο του 2018. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο είναι πιο μακριά στο μέλλον. Η αγορά των futures δεν δίνει κάτι τέτοιο. Και μετά τα F.E. δίκτυα. Από τον κομμάτι αυτού, αν θέλουμε μια αγορά όπου ε, συμμετέχει η ζήτηση, ότι δεν προσαρμόζεται μόνο η παραγωγή στη ζήτηση, αλλά και η ζήτηση στην παραγωγή και η παραγωγή μπορεί να είναι όπου θέλει και η ζήτηση όπου θέλει, χρειαζόμαστε ένα δίκτυο το οποίο είναι σε θέση να τα χειρίζεται όλα αυτά, ένα δίκτυο που μπορεί να χειριστεί σε πραγματικό χρόνο την ισορροπία που απαιτείται για να εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω τις απαντήσεις α, ανταποκρινόμενες στις σκέψεις των Ευρωβουλευτών. Αν επιτρέπετε θα ξεκινήσω από εσά και τη σκέψη για τον κατακαιρματισμό της πραγματικότητας. Δώσατε την πραγματική εικόνα. Γι' αυτό, επειδή έχουμε διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη όσον αφορά την προώθηση των ΑΠΕ και την ένταξή τους, δεν βρίσκουμε μια και μοναδική λύση που να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ούτε για τους διάφορους τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η θέρμανση, η ψήξη, η ηλεκτρική ενέργεια, ούτε όσον αφορά την ταχύτητα αναπτύξεως των δικτύων κατά τομέα σε κάθε χώρα. Εγώ το 2001 και, πέρα παρακολουθούσα τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Πάντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλαμε να έχουμε ένα αρμονισμένο μηχανισμό υποστήριξης και πολύ συχνά εμπόριο ποσοστώσεων και επιστοποιητικών. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα και εφαρμόστηκε, ελάχιστα ήταν αυτό. Ποτέ δεν έτυχε υποστηρίξει. Και δεν θα χρονοτριβούσα προσπαθώντα να κάνω κάτι παρόμοιο. Θα ήταν τόσο μικρό ο παρονομαστή που δεν θα μπορούσε να μας επιτρέψει να πετύχουμε το στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 27%. Και ερχόμαστε στον κύριο Λάγκε. Είπε ο κύριος Λάγκε πόσο χρειαζόμαστε, πόσο χρόνο χρειαζόμαστε ε, για τις τιμές ή μία τιμή θα έλεγα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μια τιμή. Δεν είναι ο ιδεώδης ο κόσμος στον οποίο ζούμε και ο ενεργειακός τομέας είναι περιπλοκότατος. Βρήθη ε, τιμών, φόρων, επιδοτήσεων, μη εσωτερικευμένων, ελάχιστα εσωτερικευμένων και κοινωνικών καθηκόντων και στόχων. Όταν οι χώρες έχουν ρυθμιζόμενες τιμές για τα α, νοικοκυριά ή για τη βιομηχανία και βγάζουν τη βιομηχανία και δεν χρειάζεται να πληρώσει το κόστος του δικτύου βιομηχανία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Γι' αυτό, αν θέλετε να κινηθείτε προς 100% σε ανανεώσιμες μέχρι το 2050 ή 50% μέχρι το 2040, τότε χρειάζεται ασφάλεια επενδύσεων. Και η τεχνολογία που έχει μόνο κόστος κεφαλαίου και όχι καθόλου κόστος, έχει μόνο πάγιο κόστος, η τράπεζα λέει, σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποιο προσθήκη για τον κίνδυνο και γίνεται η χρηματοδότηση. Και η κυρία από τη Σκανδιναβία, η Ευρωβουλευτής, είπε κάτι. Συμφωνώ δεν ήθελα να μιλήσω μόνο για την ανανεώσιμη παραγωγή από, από ανανεώσιμες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκθεσή σας αργότερα θα το τονίσει αυτό που θα πω τώρα. Υπάρχουν τομείς που δεν αντιμετωπίζονται σωστά στον κόσμο των ανανεωσίμων. Μεταφορές και θέρμανση. Πρέπει να βρούμε καλό παράδειγμα από τη Σουηδία και τη Δανία στι μεταφορέ, γιατί είναι πιο προχωρημένε από άλλε χώρε αυτέ. Θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή πρακτικών, με άλλα λόγια. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ερώτηση, γιατί η, παραμένει σταθερή και δεν χρησιμοποιείται η δυνατότητα παραγωγής στο φυσικό αέριο όταν το δίκτυο προσπαθεί να ισορροπήσει. Αυτό δεν είναι εύκολη απάντηση. Με την έμπριον στη ζώνη τη γερμανική βλέπει κανείς ότι έχουμε πολύ άνθρακα στο σύστημα ίσως είναι άνθρακας και πυρηνική. Εάν θέλετε να, να εξαλείψετε τον άνθρακα, το σκέφτεται η κυβέρνηση, άρα θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για παραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης μέσω φυσικού αερίου. Και το θέμα είναι τι κάνουμε με τα διάφορα εργαλεία ένταξης και ολοκλήρωσης. Όταν μιλάτε για, τον, για την αγορά, μου άρεσε η ιδέα του εμπορίου των διαφόρων ορίων των τιμών, αλλά μεταβάλλεται η ζήτηση και η προσφορά. Σε βιομηχανικό επίπεδο, σε επίπεδο νοικοκυριών υπάρχει αλλαγή στη ζήτηση. Υπάρχει, υπάρχουν τοπικά έργα από, από συνεταιρισμούς, από διάφορα νοικοκυριά και δημιουργούν ανάγκες που ε, ζη, απαιτεί ευελιξία για να καλυφθεί. Και για να ανταποκριθεί κανείς τευμετάβλητο χρειάζεται ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται και αυτή είναι η ομορφιά είτε στη διαχείριση του δικτύου είτε ομαδοποιώντας φορτίων από μικρές μονάδες αλλά αυτό που πραγματικά δηλητηριάζει την προσπάθεια για ευελιξία, για πλήρη ευελιξία, είναι ο μηχανισμός ισχύω με βάση το φορτίο, παλιά ιδέα. Αν δημιουργείται σε την αγορά δυναμικού θα είναι ε, κάτι το οποίο δεν είναι καλό για κανέναν. Εμποδίζει την πρόοδο. Δεν δημιουργεί καμία ασφάλεια για εκείνους που έχουν τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας. Και πάμε σε επιδοτήσεις. Συμφωνώ ότι για αλλαγή υποδομών και βιώσιμη αλλαγή της υποδομής που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη με διάφορες ταχύτητες και γενικότερα πιθανότατα αυτό θα οδηγήσει σε νέες επιδοτήσεις. Αυτό εννοούσα στις διαφάνειες που σας έδειχνα. Δεν θα πρέπει να ονειρευόμαστε. Οι παλιέ μονάδε πυρηνική ενέργεια, είτε σα αρέσει πυρηνική ενέργεια ή όχι, οι, πολύ, οι απειρχιωμένε μονάδε παραγωγή με πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να ε, ε, έχουν κλείσει από παλιά για λόγους ασφαλείας. Θα χρειαστούν πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν θα τα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάζονται χρήματα που δεν υπάρχουν για να γίνει αυτό. Στο τέλος θέλουμε ένα ασφαλή κόσμο και θα πρέπει να πληρώσουμε για την ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για υποδομές, για ενισχύσεις για τις υποδομές και για εξάλληψη του άνθρακα και της πυρηνικής και θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου και παρακαλώ εσείς τώρα. Ευχαριστώ. Μερικές από τις ερωτήσεις αφορούσαν αντίστοιχα θέματα και θα προσπαθήσω να τι ομαδοποιήσω. Η πρώτη ερώτηση του κυρίου Λάγκεν για την ε, αγορά μέσα στην ίδια μέρα intraday market. Αν μου επιτρέψετε θα το πω κάπω διαφορετικά. Η αγορά αυτή δεν είναι τμήμα του προβλήματος, είναι τμήμα της λύσης. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια ε, για να έρθει πιο κοντά στην πραγματική ζωή, στον πραγματικό χρόνο. Ε, ε, σήμερα οι αγοροπολισίες γίνονται και μισή ώρα πριν την παροχή. Στα δύο συνοριακά είναι μία ώρα αντί για μισή, γιατί χρειάζεται ευξημένη συνεργασία ιδιαίτερα μεταξύ ε, των ε, διαχειριστών και δεν είμαστε εμείς ε, σε αυτό το χώρο. Έχουμε ένα παράδειγμα γιατί πώς μπορεί η μερίσια αγορά να βοηθήσει να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την προσφορά. Το 2014 στην έκλειψη ηλίου υπήρχαν κάποιες, κάποια αποθέματα. Το είχαν προβλέψει στη Γερμανία αλλά ε, δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν ε, την έλλειψη του ηλεκτρικού ρεύματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της έκλειψης ηλίου. Άρα ακριβώς δεν υπήρξε πρόβλημα, παρόλο που ήταν μεγαλύτερη ζήτηση και μικρότερη προσφορά, ε, λόγω της ημερήσιας αυτής αγοραπολισίας κατάφεραν να καλύψουν τις ελλείψεις αγοράζοντας ρεύμα από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αλληλένδετα και έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του συστήματος. Η ημερήσια αγορά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Ε, θα πρέπει να βασίζεται σε μια πολύ ε, γερή βάση γενικότερα για την εξορρόπηση της αγοράς και θα πρέπει να αφιερωθούμε σε αυτό και να αφοσιωθούμε σε μια πιο ε, πανευρωπαϊκή προσέγγιση και να ενταχθούν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτό που σήμερα δεν υπάρχει ως δυνατότητα σύντομα δύο λόγια για τα νέα προϊόντα όπως είναι ε, συμβόλαια ενός τετάρτου της ώρας, 15 λεπτών δηλαδή, που έχουν ε, εισαχθεί, δεν ξέρω αν μπορούν να ε, γίνουν συναλλαγές και διασυνοριακές, πάντως ε, αυξήθηκαν οι συναλλαγές και βλέπουμε και να δραστηριοποιούνται και η παραγωγή ΑΠΕ. Κάτι που δεν έχει ε, ακόμα αναπτυχθεί είναι η ξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες 24 ώρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ε, από όλες τις χώρες δεν υπάρχει τόση ανάλυση ευθύνη, χρειάζονται και περισσότερα κίνητρα για να αυξηθεί η ρευστότητα. Ε, κάτι άλλο που ακούστηκε ως ενδιαφέρον σχόλιο για τον τίτλο της έκθεσης. Αν είναι ένα σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, είναι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρω ότι είναι θέμα γλωσσικό αυτό, ε, θέλω να φωτίσω ένα θέμα που δεν είναι καθόλου κρίσιμο ή επικριτικό στην έκθεση, αλλά πρέπει να τα κρατήσουμε χωριστά αυτά. Είναι διακριτά τα πράγματα. Όπως για τους στόχους του κλίματος έχουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων στην Ευρώπη που θα πρέπει να ενισχυθεί για να φτάσουμε τους στόχους μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το εντάξουμε στο σχεδιασμό της ε, ενεργειακής αγοράς. Αυτό θα αυξήσει την περιπλοκότητα. Ως ε, γενικότερη αρχή είναι καλύτερο να έχεις ένα στόχο για να αντιμετωπίζεις ένα ζήτημα τη φορά. Έγιναν και άλλες ερωτήσεις για τις αγορές ισχύως ε, capacity markets. Ίσως επικρατεί κάποια σύγχυση για το τι σημαίνει αυτό και περί τίνος πρόκειται. Capacity mechanisms markets ή επιδοτήσεις ή συστήματα υποστήριξης επιδοτήσεων να προσπαθήσω λίγο να βάλω μια τάξη. Και από τη δική μας σκοπιά είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το εξής. Οποιοδήποτε σχεδιασμός αγοράς ε, για να σταθεί στο μέλλον θα πρέπει να ανταμείβει και την ισχύ σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, αυτό στην αγορά ενέργειας είναι πολύ σαφές, ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως ο σχεδιασμός της αγοράς όπως είναι σήμερα έχει τέτοια στοιχεία. Όπως είναι η αγορά εξισορρόπησης που κυριαρχεί όταν υπάρχει μειωμένη ε, ε, ισχύς και, και αμείβεται η παραγωγή της. Υπάρχουν λύσεις και σήμερα δηλαδή και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Ε, ίσως χρειάζεται να αναπτυχθούν περισσότερο. Ακούστηκε και αυτό προηγουμένως. Η υποστήριξη χρηματοδοτική και επιδότηση των ανανεωσίμων σε κάποια κράτη ακριβώς τονώνουν και τις επενδύσεις ε, στην ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα και στην ισχύ, τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μεταφράζεται σε παραγωγή ενέργειας, υπάρχουν πάντως μηχανισμοί στήριξης της παραγωγής. Αυτό που δεν χρειάζεται επιπλέον είναι νέες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, ιδιαίτερα όταν ε, μπαίνουν ε, και επηρεάζουν τη τιμολόγηση. Για λόγους πολιτικούς ή οικονομικούς, όποιους λόγους και να έχει ο καθένας, πάντα μπορεί να αξίζει να υποστηρίζει κάποιες τεχνολογίες ε, ελπιδοφόρες, καινοτόμες ως πιλωτικά προγράμματα για να μπουν στην αγορά και να αποκτήσουν ε, ανταγωνιστικότητα και ε, ώστε να μην χρειάζονται στο μέλλον οικονομική υποστήριξη. Πάντα γίνεται αυτό, αλλά χωρίς να στρεβλώνει την αγορά energy only. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πληρώνει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, να επιδοτείται στο βαθμό ε, που δεν μπορεί να καλύψει το κόστος του μέχρι να μπορεί να ε, κερδίζει τόσα πολλά από την παραγωγή και την κυκλοφορία στο δίκτυο της αγοράς, ώστε να μην χρειάζεται επιδότηση. Αυτό χρειάζεται εκ των υστέρων ε, αξιολόγηση και να αντιμετωπιστούν και κάποιες ελλείψεις από τη μη βέλτιστη συμμετοχή στην αγορά. Δεν θα πρέπει να επιδοτούνται δηλαδή ζημιογόνοι παραγωγή. Δεν υπάρχει ουσιαστικά πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάποιες συμβατικές τεχνολογίες. Μπορεί να υπάρχουν και πολύ ευέλικτε ε, συμβατικές τεχνολογίες που αξίζει να υποστηρικτούν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με ακριβώ τον ίδιο τρόπο μέχρι να σταθούν στα πόδια του ε, ε, βαρός και πριν μπουν στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας και τους τρεις ομιλητές του πάνελ αυτού. Πάρα πολύ ε, ενημερωτικά αυτά που μας είπατε, περιστατωμένα, εκτενής προσέγγιση και συνολική και σφαιρική. Ε, μεγάλο χειροκρότημα σας αξίζει και να τα ξαναπούμε στην Επιτροπή. Uh, Ο πρόεδρος Μπούσεκ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το δεύτερο πάνελ. Διαχειριστές, διαχειριστές ε, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και ρυθμιστές. Πρώτος ομιλητής τώρα, ο κύριος Πέντερ Όστερμαρκ Άντρεασεν. Ο κύριος Αντρεάσεν που είναι εκλεγμένος πρόεδρος της E του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταδόσεως. Και ως γνωρίζουμε είστε και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EnergyNet Ζουδανίας. Και είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Ένωσης ε, ε, παραγών του ρεύματος Δανία. Δεν έχετε πολλούς παραγωγού, έχετε πολλούς χρήστε και ρυθμιστές. Αυτό είναι ενδιαφέρον για μας και θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε τι έχετε να μας πείτε. Διότι για το σχεδιασμό μάλλον τη αγορά ηλεκτρικής ενέργεια. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω ότι ο διάλογος μεταξύ ευρωβουλευτών και του κλάδου μας είναι ε, πολύ σημαντικός και γόνιμος. Θα ανεφερθώ σήμερα στην ε, άποψη του Έντσο Ι. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν για την έκθεσή του βεβαίως και θα επανέλθω προς το τέλος για να ε, μιλήσω για την έκθεσή σας. οι TSO, οι διαχειριστές δηλαδή συστημάτων, είμαστε ικανοποιημένοι από την COP21 γιατί μας δίνει ένα ξεκάθαρο δικό χάρτη. Ξέρουμε ότι μέχρι το 2030 θα χρειαστεί να έχουμε πάνω από 45% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ε, σύστημα. Το μέγα ερώτημα είναι, είναι δυνατό να γίνει αυτό. Δεύτερο, είναι δυνατό να πληρωθεί νομίζω ότι από την έντσο μπορούμε εμείς να πούμε ναι εφόσον γίνει με σωστό τρόπο. Είναι σωστές επίσης οι θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς θα αναπτύξουμε τις αγορές και τους στόχους υποδομών. Ένα από τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για να φτάσουμε στο 45% ίσως και 50% των ανανεώσιμων είναι η ευκαμψία. Έχω εδώ ένα χάρτη που σας δείχνει τις ανάγκες αυτές. Πρόκειται για μια εβδομάδα παραγωγής ενέργειας στην Δανία. Έχετε τις γκρίζες ε, ζώνες που κατανάλωση και το γαλάζιο που είναι ε, ηλιακή ενέργεια και αιωλική ενέργεια. Γι' αυτό μιλούμε και για ευκαμψία. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό στην ε, Δανία, συμβαίνει όμως και σε πολλές άλλες περιφέρειες. Και στη Γερμανία μπορεί να είναι και χειρότερο από το, την εικόνα που βλέπετε εδώ. Άρα χρειαζόμαστε ευκαμψία όχι μόνο του συστήματος, αλλά και από τους διαχειριστές των συστημάτων διανομής. Γιατί η περισσότερη από την ενέργεια αυτή, ηλιακή και αιωλική, πηγαίνει στο δίκτυο διανομής. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν ε, ανάγκες ε, ελέγχων. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας για να προχωρήσουμε. Θέλουμε λοιπόν, όπως είπα, περισσότερη ευκαμψία για να μπορέσουμε να περιλάβουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα. Το βασικό μας μήνυμα είναι ότι θέλουμε να μειωθεί η κατά διανομή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε έξω τις ανανεώσιμες. Αντίθετα, να μπορέσουμε να βάλουμε στο σύστημά μας πολύ περισσότερες ε, ε, ανανεώσιμες εάν σταδιακά καταργήσουμε το priority dispatch. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως για την κατάργηση της ε, κατά προτεραιότητα πρόσβασης, διότι οι ανανεώσιμες έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση γιατί έχουν κόστος σχεδόν μηδέν δηλαδή για την ε, αγορά της επόμενης ημέρας θα έχουν σχεδόν αυτομάτως ε, ε, προτεραιότητα. Δηλαδή θα είναι οι πρώτες που θα εξυπηρετηθούν στην αγορά και έχουμε ηλιακή και ολική σχεδόν 50% στη Δανία και πολύ σπάνια τις περιορίζουμε παρόλο που δεν έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση αλλά λόγω του σχεδιασμού της αγοράς θα εξυπηρετούνται πρώτες. Βέβαια, όταν οι τιμές είναι αρνητικές θα πρέπει να σταματάμε τις ανεμογεννήτριες αν δεν έχουμε επαρκή υποδομή για να επιτρέψουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αλλά εδώ δεν μιλούμε μόνο για τις ανανεώσιμες, εδώ μιλούμε για το σχεδιασμό της αγοράς στο σύνολό της. Οι ιδέες που έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις ιδέες της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου είναι θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της αγοράς πρέπει να στραφεί γύρω από κύκλους που θα αντιμετωπίζουν τη σπάνιδα των ε, πηγών. Σε ένα ειδόδι κόσμο θα λέγατε ότι η τιμή του προϊόντος απηχεί όλα τα χαρακτηριστικά του. Όταν μιλάμε όμως για την τιμή προϊόντος του ηλεκτρικού ρεύματος, το μόνο που περιλαμβάνει είναι το κόστος που έχει απήξει την αγορά. Πρέπει να δείχνει και την ευκαμψία. Πρέπει η τιμή δηλαδή να περιλάβει και το κόστος ευκαμψίας. Και χρειαζόμαστε περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα για να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη ευκαμψίας και σπάνιδος. Αυτό θα μας απασχολήσει. Περισσότερη αγορά. Ώστε να μπει τιμή, μια σωστή τιμή πάνω στην ευκαμψία που χρειαζόμαστε. Εμείς δεν βλέπουμε μεγάλη ανάγκη για capacity markets, βλέπουμε όμως ανάγκη για αγορά ευκαμψίας που είναι μεγαλύτερη ανάγκη από την capacity, από το δυναμικό. Και γι' αυτό ζητούμε και στενή συνεργασία μεταξύ TSO και DSO σε όλες τις ε, πτυχές της αγοράς. Συμπεράσματα τώρα από το σχέδιο εκθέσεως του κύριου Λάγκεν. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συστάσεις σας αγαπητέ Λάγκεν διότι ανταποκρίνονται και στην ανάλυση που κάνουμε και εμείς. Ένα από αυτά που προτείνουμε εμείς και το περιλαμβάνετε και εσείς στην εκθέση σας κύριε Λάγκεν είναι ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία για να κάνουμε την ανάλυση επάρκειας των συστημάτων, όχι μόνο αναχώρα, αλλά και στο περιφερειακό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΝΤΣΟΗ έχει αναπτύξει ένα σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο και ευχαρίστω να προτείνουμε να μπει, να ενταχθεί στη μελλοντική νομοθεσία. Ένα από τα πράγματα που απαιτούνται επίσης για περισσότερες αναλογισμένες ενέργειες σημαίνει και περισσότερη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και μεταξύ TSO. Εμείς συνεργαζόμαστε εδώ και 100 χρόνια, ε, TSO δηλαδή, διαμεθοριακά. Έχουμε ιστορία πολύ μακρύτερη από τη ίδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ένωσης, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία. Και γι' αυτό αναλαμβάνουμε πολλές πρωτοβουλίες συνεργασίας για να ενισχύσουμε το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή. Και των όσων εφαρμόζουμε τώρα, αλλά και για να φτιάξουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να ενσωματωθούν, να ενταχθούν όλες αυτές οι ανανεώσιμες στα συστήματα. Η δε τελική ευθύνη για την ασφάλεια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θα βαρύνει εν τέλει τους τοπικούς TSO και τις τοπικές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η TSO δεν είμαστε ένα ελεύθερο άτομο το οποίο ε, κυμαίνεται στα εθέρια στρώματα, αλλά εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική στήριξη και από τη ρυθμιστική στήριξη. Το έχουμε αυτό στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στις χώρες μας. Για να μπούμε τώρα στην περιφερειακή φάση πρέπει να δούμε να αναπτύσσεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο που να εξυπηρετεί αυτή την περιφερειακή συνεργασία. Αυτή είναι η έντονη επιθυμία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι τοπικές αυτοδιοίκησεις να μπορέσουν να μας δώσουν αυτή την πολιτική στήριξη. Τα είδαμε αυτά στα πρώτα βήματα της συνεργασίας και μπορούν να ενισχυθούν. Μας ικανοποιεί η πρότασή σας για την ενίσχυση της Acer. Όντως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη και μάλιστα περισσότερη στήριξη δηλαδή. Το ίδιο η αποτελεσματική στήριξη των εντολών, των φυστραμένων εντολών για την ΕΣΕΡ και το ΕΝΤΣΟΗ e, για να υπάρξει ευκαμψία της διανομής στο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το πολύ ξεκάθαρο και έντονο μήνυμά σας προς όλες και όλους μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως. Μήνυμα το οποίο βρήκα πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια πάντα είναι πιο εύκολο για μας με τα μήνυματα αυτά να κατανοήσουμε καλύτερα το όλο θέμα. Ο κ. Ντόναλντ Βαν Μπέβερεν, διευθυντής ρυθμιστικών του βελγικού συστήματος διανομής. Που λειτουργεί στη Φλάνδρα και παρέχει λύσεις δικτύου για, ε, για τη δημόσιο φωτισμό, ηλεκτροδότηση, φυσικό αέριο. Θα κάνει την παρέμβαση. Ο κ. Βαν Μπέβερεν είναι πολιτικός μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την ευκαιρία που μας δίνετε να έρθουμε να σας δώσουμε την άποψή μας ως διαχειριστής του δικτύου. Εγώ θα μιλήσω για τις ε, προκλήσεις πρώτα, μετά για τις λύσεις και κάποια παραδείγματα και μετά σε ποιο βαθμό ε, αυτό αφορά τον τελικό καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις αυτές, ε, βεβαίως ε, ακούσαμε από όλους τους ομιλητές ποιες είναι αυτές, ε, ανανεώσιμες, αποκέντρωση, ηλεκτροδότηση, εξηλεκτρισμός, ξεκάθαρα όλα αυτά. Ως λοιπόν δι, διαχειριστής του δικτύου έχουμε πάρα πολύ προσαρμόσει τις δραστηριότητές μας, έχουμε δώσει και εφαρμόσει κάποιες τεχνικές λύσεις και τεχνολογικές και εκτός αυτού ε, είμαστε πλήρως αποσυνδεδεμένοι. Εγώ βέβαια είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω εγώ για το Βέλγιο, ε, ότι είμαστε πάντα οι καλύτεροι μαθητές ε, στην ευρωπαϊκή τάξη, σε καμία περίπτωση, αλλά για την αποσύνδεση είμαστε πραγματικά άριστοι μαθητές. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι το δίκτυο στην Ευρώπη διαφέρει πάρα πολύ για τους διαχειριστές και ε, στο θέμα της, του μεγέθους του δικτύου, το διαχειριστή, την αποσύνδεση και ε, αν τα δίκτυα είναι ήδη ευφύ ή όχι. Όλα αυτά είναι πράγματα που διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα και μάλιστα από περιφέρεια σε περιφέρεια θα έλεγα. Τώρα, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης γίνεται λόγος για το ρόλο του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς που αλλάζει επίσης. Ε, κάποιες δραστηριότητες, κάποια νέα καθήκοντα αποκτούμε, αλλά και ένα νέο ρόλο. Ε, σας έχω εδώ επισημάνει ορισμένα ε, ένας ουδέτερος διευκολυντής πρόσβαση στην αγορά, ενεργειακή απόδοση, εφείς μετρητές, η διαχείριση δεδομένων. Και αυτό που έχει σημασία είναι η αποθήκευση σε συσσωρευτές, σε μπαταρίες ως τεχνική λύση. Αν καθίσουμε να σκεφτούμε τι γίνεται και πώς μπορεί όλες αυτές οι δραστηριότητες να αφορούν ένα διαχειριστή δικτύου μεταφοράς. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι. Ε, και ανάλογα με το αν είναι αποσυνδεδεμένος ή όχι και σε ποιο βαθμό διαχειριστής, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανεξαρτησία και για ουδετερότητα. Αν θέλουμε να γνωρίσουμε ένα ρόλο στο διαχειριστή, υπάρχουν βεβαίως πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα. Ποια είναι τα υπέρ. Ε, μπορεί πιο γρήγορα να αναπτυχθεί η αγορά, μπορεί να λυθούν κάποια προβλήματα για το ποιο έκανε πρώτο η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Υπάρχουν μερικά προβλήματα που έχουν οι ε, νεοφύης επιχειρήσεις σχετικά. Ε, άλλο πλεονέκτημα είναι η ομοιομορφία και η διαλειτουργικότητα των λύσεων. Υπάρχουν ενδεχομένως και ε, τα κατά που βλέπετε εδώ σε αυτό το πίνακα. Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής, τις δραστηριότητε, τι γίνεται με την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τι γίνεται με την καινοτομία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Καταρχάς πιστεύουμε και εμείς ότι τα μειονεκτήματα μειώνονται δραστικά ως προς τον αντίκτυπό τους στο βαθμό που είμαστε αποσυνδεδεμένοι ως διαχειριστές του δικτύου μεταφοράς. Και ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας, δηλαδή με δύο λόγια πώς μπορούμε να μειώσουμε τα μειονεκτήματα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι και το κάνουμε κιόλα και δραστηριοποιούμεθα ε, για να ε, ε ξεκαθαρίσουμε ε, το πεδίο εφαρμογή, να ξέρουμε ποιες είναι οι δραστηριότητές μας και έχουμε και δείκτες επιδόσεων και μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να μετράει τις επιδόσεις και επίση, και δεν χωρά καμία αμφιβολία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ε, για καινοτομία μέσω εμπορικών φορέων. Και το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Θέλω να σας παραπέμψω λίγο σε κάτι που είπε ο προλαλής σας σήμερα στο Βέλγιο ως διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς και εν και της ενεργειακής μετάβασης ε, δεν έχουμε καμία ενθάρρυνση για καινοτομία και για επένδυση στα ευφυή e δίκτυα. Το κάνουμε παρόλα αυτά χωρίς να έχουμε στήριξη. Επίσης σας είπα ότι ε, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα ε, από τα όσα κάνουμε σήμερα, δύο παραδείγματα διαχειριζόμαστε το δίκτυο μεταφοράς στο Γαλλίο και δημιουργούμε τώρα ένα clearing house, ε, για ε, ένα data hub για να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα αυτή για να δούμε τι γίνεται στο δίκτυο μεταφοράς. Το χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς της αγοράς αυτό πλατφόρμα αγοράς και ε, στη δομή διακυβέρνησης αυτού που ονομάζεται Άτριας, αυτή η οργάνωση που συστήσαμε, συμμετέχουν και οι εμπορικοί φορείς όπως είπαμε, όπως και ο διαχειριστής και ο ρυθμιστής. Δηλαδή, πώς το λένε αυτό με το only, δεν είναι stand alone εν πάση περιπτώσει των ε, διανομέων, αλλά ε, είναι και οι διαχειριστές του δικτύου που επενδύουν. Δεύτερο παράδειγμα, ε, υπάρχει αγορά ευέλικτη στο Βέλγιο και στη διανομή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ε, για τα νοικοκυριά απέχουμε πόρο, αλλά για τη βιομηχανία πραγματικά υπάρχει ευκαψία και ευελιξία για τους πελάτες και τι ρόλο διαδραματίζουμε εμείς, το ρόλο του ε, ανεξάρτητου διαχειριστή δεδομένων και του ουδέτερου διευκολυντή της αγοράς. Από την άλλη, διευκολύνουμε ακριβώς την αγορά ευελιξίας και τα προϊόντα του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς που είναι η παραγωγή, οι προμηθευτές, ε, εκείνοι που ενοποιούν την παραγωγή και τη συγκεντρώνουν και φροντίζουν να λειτουργεί καλά. Εμείς τους δίνουμε μια πλατφόρμα, τους προσφέρουμε αυτό το εργαλείο για να διευκολύνουμε, αλλά δεν συμμετέχουμε οι ίδιοι σε αυτή την προσπατέλωση. Τι γίνεται με τον τελικό καταναλωτή, γιατί γι' αυτόν τα κάνουμε όλα αυτά. Ε, εμείς ως διαχειριστές της διανομής ε, θέλουμε να υπάρχει ενεργειακή απόδοση επίσης. Ε, διευκολύνουμε και τη σύνδεση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καμιά φορά μπορούμε να βοηθήσουμε ε, για να μειωθεί το πικ της κατανάλωσης αλλά και ο όγκος ε, που χρησιμοποιεί. Βεβαίω, πέρα από αυτό, έχει τη δυνατότητα ελεύθερο καταναλωτή να επιλέγει τον προμηθευτή του και να αλλάζει. Ε, και ε, στο επίπεδο της βιομηχανίας και εκείνο που συγκεντρώνει ε, τη παραγωγή και το, το ΕΣΚΟ που είναι η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες για την ενέργεια. Επίσης μπορεί να επιλέγει το τύπο συμβολέου που θέλει και να συμμετέχει στην αγορά ευελιξίας και σε επίπεδο διανομής και δικτύου. Και τέλος ο πελάτης μπορεί να συμμετέχει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ε, σπάνιδος ή έλλειψης μπορεί να συμμετέχει με μείωση της ίδιας του της πρόσβασης στο δίκτυο για να βοηθήσει με λιγότερη κατανάλωση να μην επιβαρύνεται το δίκτυο. Αυτά σύντομα είναι οι θέσεις που θέλαμε να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Επόμενος ομιλητής, Dr. Anne Grable, επικεφαλής του τμήματος για την, το συντονισμό για το δίκτυο ε, ηλεκτρισμού ε, ταχυδρομείων, σιδηροδρόμων, φυσικού αερίου κλπ. Πάρα πολλά θέματα καλύπτονται και είσαστε και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών Δικτύων και μέλος της ΆΣΕΡ του Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών. Άρα είναι η άποψη των ρυθμιστικών φορέων. Άλλη θέση από εκείνους που χρησιμοποιούν τα δίκτυα. Οι εκπροσωπή των ρυθμιστικών αρχών. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν τις ε, απόψεις σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά που προσκαλέσατε και τον ρυθμιστή. Θα μιλήσω στα γερμανικά διότι ε, νομίζω ότι έχω προσκληθεί εκ μέρους του ε, γερμανού ρυθμιστού και γιατί θα μιλήσω για την συνεργασία και συντονισμό των ρυθμιστών ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνουν και οι διάφοροι ρόλοι μου. Και θέλω πρώτα να πω ότι είναι σημαντικό να δει κανείς την αφετηρία από την οποία έχουμε δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Η αφετηρία αυτή είναι δυσχερής διότι οι χώρες μέλη στο εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με το άρθρο 149 έχουν την ευθύνη για το ενεργειακό μείγμα ενέργειας σε όλε τις ευρωπαϊκές λύσει πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Δηλαδή πάντοτε χρειάζεται να διατηρούμε μια ισορροπία, να αποκαθιστούμε μια ισορροπία μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων λύσεων. Και μάλιστα αυτές οι οποίες έχουν προταθεί. ποιε είναι, είναι τα δύο αυτά καθήκοντα. Αφενός βέβαια η ένταξη των ανανεώσιμων στην αγορά, στο εμπόριο, στα δίκτυα που ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καταφέρουμε και που απαιτεί κάποιες προσαρμογές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης η ε, ολοκλήρωση, δηλαδή η ευρωπαϊκή, ενέργεια, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε από κοινού ταυτοχρόνως και τότε θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, να μην μένουν δηλαδή σε ανταγωνισμό, τα μένουν προς τα δε. Αυτό είναι ουσιώδες ουσιώδες ως αφετηρία για τις σκέψεις που έχω να σας αναπτύξω. Και κατά τα λοιπά θεωρώ ότι η καλύτερη απόπειρα λύσεως θα είναι εκείνη που προτείνουμε ως οργανισμός, ομοσπονδιακός οργανισμός για τα δίκτυα και παρακολουθούμε τώρα στην Ομοσπονδιακή Γερμανία μια αφετηρία μιας αγοράς energy only και κρίσιμο εδώ για να λειτουργήσει αυτή η λύση στη βάση της αγοράς και τα μηνύματα που θα δίνουν οι τιμές να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα είναι πρώτα-πρώτα να τους αφήσουμε στην ισχύα τους. Δηλαδή να μπορέσουν να εργαστούν χωρίς τρευλώσεις. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τροποποιηθούν οι μακροπρόθεσμες συνθήκες πλαίσια για να έχουμε μετά πάλι την σύμπτωση των όσων σήμερα ξεφεύγουν από ένα κοινό πλαίσιο, δηλαδή των μακροπρόθεσμων αναγκών σε επενδύσεις που όμως δεν είναι δυνατό να λυθεί με νέες επιδοτήσεις, με capacity markets και το καθεξής. Πρέπει να λυθεί αφήνοντας να περάσουν μηνύματα μιας ε, άνευστρεβλώσεων αγοράς. Αυτό καθίσταται σαφές στην έκθεση και αυτή είναι και η δική μας αντίληψη. Αυτό σημαίνει εξάλλου, όπως είπα προηγουμένως, δεν θεωρούμε αναγκαίες τις ε, capacity markets. Αυτό σημαίνει ότι μετά από μια μεταβατική φάση και από την πλευρά των ε, ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας πρέπει να δώσουμε κάποια οικονομικά κίνητρα για να συμπεριφερθούν με τρόπους προσαρμοσμένους στην αγορά. Αυτή η εξέλιξη έχει ήδη αρχίσει, έτσι νομίζω. Η αρχική δηλαδή φιλοσοφία, η οποία ασφαλώς ήταν αναγκαία για να προωθηθούν οι ανανεώσιμες ενέργειες και η οποία απέληξε σε ένα είδος φιλοσοφίας produce and forget έχει ξεχαστεί πλέον και στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Και είναι σκόπιμο, όπως είπα, να οδηγηθούμε σε ανευστρεβλώσεων οικονομικές συμπεριφορές. Και τότε θα λειτουργήσει η energy only αγορά. Και ασφαλώς πλέον μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αναλυφθεί μια ευθύνη των οικονομικών κύκλων για την για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία με τη μεταρρύθμιση του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε περιλάβει περισσότερα στοιχεία αγοράς στη νομοθετική αυτή ρύθμιση για να προκαλέσουμε την συμπεριφορά αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει ακόμα η κατά πρόσβαση, priority access, αλλά και εδώ είναι καθαρό ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει επάπειρον. Και εν τέλει όλα τα στοιχεία της αγοράς θα πρέπει να μπορούν να δρουν και να λειτουργούν χωρίς τρευλώσεις. Ιδάλλως δεν πρόκειται να λειτουργήσει η βασική αρχή του μηχανισμού ε, της, ε, που βασίζεται στην αγορά. Για να το απηχήσουμε αυτό, είναι σωστό αυτό που λέχθηκε ήδη από τον προλαλήσαντα, ότι δηλαδή είναι ένα σημαντικό στοιχείο ότι η ευκαμψία θα πρέπει και αυτή ε, να ε, επιτραπεί και όχι μόνο από στην πλευρά του balancing και αυτό δεν δέχθηκε απόλυτα καθαρά ιδίως και από την πλευρά της ζήτησης demand side responsibility εκεί θα αποτελέσει ένα κέριο στοιχείο και μάλιστα στοιχείο το οποίο είναι δύσκολο να εισαχθεί διότι έχουμε διαφορετικές ομάδες ζήτησης και πρέπει να δούμε εκεί πώς θα λειτουργήσουν στην αγορά. Μου φάνηκε σημαντικό ότι από το χρηματιστήριο ήδη έχουν εισαχθεί ορισμένα προϊόντα στην πλευρά αυτή που καθιστούν δυνατή την, ε, ε, την εξέλιξη αυτή και νομίζω μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα αντιστοιχούν με τα σινιάλα και θα αναπτύσσουν αυτά τα spread, σε εύρος δηλαδή, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Μίλησα περισσότερο για το εμπόριο τώρα. Θέλω λοιπόν να αναφέρω ακόμη και εκεί στην βάση οι ρυθμιστές είναι αρμόδιοι, ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μια καλά ανεπτυγμένη υποδομή δικτύων. Και αυτή η υποδομή δικτύων πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που σημειώνονται στην πλευρά των παραγωγών. Έχουμε εδώ το εργαλείο του σχεδιασμού ανάπτυξης δικτύων με ορίζοντα δεκαετίας, ειδικά δε στην Ομοσπονδιακή Γερμανία από την ε, εποχή της αλλαγής στην ενέργεια, ενεργή Δουλεύουμε πάνω στο άνοιγμα νέων επενδύσεων σε δίκτυα για να μπορεί να ανταποκρίνεται η εξέλιξη αυτή στις αλλαγές που έχουν γίνει από την πλευρά των παραγωγών. Κάτι που είχε υποτιμηθεί αρχικά, ότι δηλαδή η δικτυακή υποδομή πρέπει να παρακολουθεί τις αλλαγές στις δομές των παραγωγών. Κέριο καθήκον βέβαια των ρυθμιστικών αρχών. Και αυτό ισχύει όχι μονάχα στο εθνικό επίπεδο, αλλά και ιδίω στην διαμεθοριακή λογική, όπου εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε εχμές και στα interconnectors. Υπάρχουν εργαλεία εδώ, υπάρχουν μηχανισμοί που με συμμετοχή των ρυθμιστών, για παράδειγμα projects of common interest, ελκύουν την προσοχή των ρυθμιστών και υπάρχουν εκεί μάλιστα και ιδιαίτερα ρυθμιστικά κίνητρα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, διαμεθοριακή κατανομή κόστους, cost water cost allocation. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτό, διότι ανοίγει την δυνατότητα κατανομής του κόστους διαμεθοριακά. Κάτι που γίνεται αντικείμενο ρύθμισης ή συντονισμού από την Acer, αλλά εφαρμόζεται πλέον από τους εθνικούς ρυθμιστές. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να θέσω τώρα στο τέλος. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη συντονισμού στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω του στοιχείου των περιφερειών. Το ακούσαμε ήδη αυτό και όντως αποτελεί ένα μέγα μέρος της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κρίσιμο εδώ είναι ο συντονισμός αυτός να είναι να έχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εθνικούς ρυθμιστές και στον οργανισμό, agency. Δηλαδή πρέπει να δει κανείς εδώ και τις δύο πλευρές. Οι ρυθμιστές διαθέτουν ένα μεγάλο μέρος μέσω των ε, ε, ομάδων εργασίας, μέσω των Board of Regulators, στο οποίο συμμετέχω ως μέλος. Έχουν ένα ρόλο λοιπόν σημαντικό σε μια διάσταση περιφερειακή ή και υπερπεριφερειακή. Άρα κατά τούτο λέω ναι, να ενισχυθεί η ΕΣΑ, ταυτόχρονα όμως και το σύστημα των ελέγχων και ισορροπιών, checks and balances, μεταξύ οργανισμού και εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Διότι η βάση της ΕΣΑ, που είναι ο οργανισμός και αποτελεί μια πλατφόρμα των ρυθμιστών για την συμπλήρωση των καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστών θα λειτουργήσει μόνο εφόσον η ανταλλαγή μεταξύ εθνικού επίπεδου και ευρωπαϊκού επίπεδου λειτουργήσει πραγματικά μέσα στα πλαίσια της ΕΣΑ. ΕΕ Αυτό προτείνει, ε, προϋποθέτει όμως ένα governance system όπου θα παίζουν τον αντίστοιχο ρόλο οι ρυθμιστές και θα έχουν το δικαίωμα συναπόφασης. Κάθε ενίσχυση του ΕΣΑ για παράδειγμα για τη ρύθμιση των new entities που βλέπουμε, θα πρέπει να ανταποκρίνεται, θα πρέπει να έχει δηλαδή από την άλλη μεριά την ε, κατάλληλη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας του ΕΣΑ. Ήταν αυτό μια τελευταία βασική πτυχή που ήθελα να ε, θέσω και με συγχωρείτε που ίσως κάπως μακρύβωρησα. Δεν πειράζει, σε ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ο εισηγητής σας πάρει το λόγο. Ήθελα να ευχαριστήσω ε, ειλικρινά για τα ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Μετά το πρώτο πάνελ μας φέρετε μια καινούργια τελείως εστίαση και παρουσίαση. Πρώτη ερώτηση προς τον πρόεδρο Ανδρέασεν και έχει ως εξής. Ποιες μορφές ε, συνεργασίας, ξέρουμε το πεταμερές ε, φόρουμ της NTSO, ε, για τους διαχειριστές των δικτύων, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία. Εσείς ε, μαζί με 40, αν δεν απατώ με επιχειρήσει συνεργάζεστε και πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. δεύτερο, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται λόγος για ε, την διαθεσιμότητα των ε, δεδομένων. Χρειάζονται οι διαχειριστές των δικτύων τα δεδομένα αυτά ή έχει δίκιο ο κύριος Βαμπέρεν που λέει ότι σε, επίπεδο DSO μπορεί, μπορεί να γίνει αυτό, όχι TSO για την ασφάλεια ε, και την ευελιξία του πελάτη. Και μια άλλη ερώτηση προς τον κύριο Βαν Πολύ ενδιαφέρον το σύστημά σας στο Βέλγιο. Ε, σε ποιο βαθμό ανατρέχουν σε αυτό ε, οι πελάτες, το αποδέχονται, έχετε μια ενδιάμεση αξιολόγησή του. Και μια ερώτηση προς την ε, κυρία δόκτωρα Κέλμπελ. Εδώ στο Κοινοβούλιο βεβαίως θα μας απασχολήσει και το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο ρυθμιστή Acer. Και θέλω να σας ρωτήσω, συντονισμός τυποποίηση ε, πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πια, πέρα από τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Τι θα πρέπει να εκχωρηθεί στον ΕΣΕΡ. Ευχαριστώ. Τώρα. Η κυρία Κομπολανάτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατη και απλούστατη. Δεν ξέρω ένα απλή και απάντηση. Ποιο επίπεδο είναι το καλύτερο επίπεδο ευκαμψίας για το σύστημα. Ίσως υπάρχει και κάποια καινοτομία για όλο το σύστημα. Θέλουμε να εξυπηρετούμε θα όταν, ότι υπάρχει ανάγκη και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, όταν δεν υπάρχει άνεμος. Στη Φιλανδία έχουμε 100%, καλύψη 60 λεπτά με τα μέτρα με τους μετρητές, δεν ξέρω στο Βέλγιο 100% περίπου. Τι γίνεται, επειδή κάναμε, εφαρμόσαμε τα νέα μέτρα πρώτη θα υποφέρουμε. Λοιπόν, ευκαμψία και αποθήκευση. Δεν θα είναι αποτελεσματική αποθήκευση όσον αφορά το κόστος ακόμα. Για την ευκαμψία υπάρχουν συστήματα που μπορούν να προσαρμοστούν σε 10 λεπτά. Ε, να αντιδράσουν με οποιοδήποτε κάψιμο τάχιστα χρειάζεται και καλή τιμή για την ευκαμψία. Σε επίπεδο παραγωγού, ο πάροχος πρέπει να εξισορροπεί τις ανισορροπίες σε επίπεδο DSO που θα τοποθετηθεί στο σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταλίτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ εκ νέου. Και τα δύο πάνελ μα αποτελούν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης δεν ξέρω αν είναι επιλογή που κάνατε. Είμαστε τυχεροί ή κατανοήσαμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά την αγορά. Ζήτω. Συγγνώμη, μόλις τελειώσει την παρέμβαση πρέπει να αποχωρήσω. Πρέπει να επιστρέψω στην πατρίδα μου, όμως οι συνάδελφοι παρακολουθήσουν τη συνέχεια της συνεδριάς και τις απαντήσεις. Καταρχήν, αυτό που είπε και ο Σαντρέασεν θέλω να θίξω και που διαφωνεί με το προηγούμενο πάνελ για την πρόσβαση προτεραιότητας. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Κύριε Αντρέασον, από ό,τι θυμάμαι, αναφερθήκατε σε πολιτική υποστήριξη στο TSO. Το αποκωδικοποιείτε σας παρακαλώ. Πώς το εννοείτε. Για την αύξηση της ισχύω του δυναμικού και για αναθεώρηση της εντολής δεν ήσασταν ακριβείς. Αναθεώρηση της εντολής που εδόθη στην Acer. Τι έχετε υπόψη, τι εννοείτε. Και σας κυρία μου, μια άλλη ερώτηση έχω. Είπατε ότι αν ισχυθεί η Acer θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πτυχή της διακυβερνήσεως παράλληλα. Δεν το αμφισβητώ. Θα εξηγούσα τη διαφοροποίησή ω όσον αφορά τον χρονισμό, αν είχαμε χρόνο. Εσείς θέλατε παράλληλη κίνηση. Εγώ θα έλεγα ότι όταν προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αγοράς, κάτι που θα πρέπει να γίνει κυρίως από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τότε και τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν επί του όλου ζητήματος. Μπορείτε να δώσετε λεπτομέρειες. Όπως είπε και ο κ. Λάγκεν, και εγώ έχω μια ερώτηση. πάμε προς ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών. Τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια στοιχεία πρέπει να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι των όσων γίνονται σε εθνικό επίπεδο και αποχωρώ. Ο κ. Σαουτάκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς αξιολογείτε τις εγκαταστάσεις της υπεράκτης offshore, τις αιωλικές. Έχουμε το πρόβλημα των διακυμάνσεων κατέρικα της ημέρας και της διασύνδεσης με τα δίκτυα. Υπάρχουν προγράμματα όσον αφορά τις υπεράκτιες αιωλικές εγκαταστάσεις μέσω υποθαλασσίων καλωδίων κλπ. Πώς το βλέπετε εσείς. Πώς τα βλέπετε αυτά τα έργα, τι πρόπτικες υπάρχουν και πώς θα επηρεαστεί η αγορά. Θα γίνεται διεθνής, ε, διεθνοποίηση των ανανεωσίμων έτσι, ομαδοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες. Και για κάποιες κυβερνήσεις ίσως αυτό να είναι προβληματικό. Ποια είναι η απόψη σας. Και εγώ έχω μια ερώτηση, λέω κύριος Μπούζεκ. Στο μέλλον, τους βρόχους μπορούμε να τους αποφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι η τελευταία ερώτηση που σας απευθύνω. Αν έχετε την καλοσύνη, αρχίστε να δίνετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Πολύ καλές ερωτήσεις. Κύριε Λάγκεν, τι είδους συνεργασίας μπορούμε να φανταστούμε για να προχωρήσουμε. Είναι ακρογωνίως λίθος για τη μελλοντική νομοθεσία αυτός, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εθνική συνεργασία πρέπει να αυξηθεί. Και πολύ μάλιστα. δημιουργούμε 5-6 περιφέρειες στην Ευρώπη για να εξυπηρετούνται περισσότερες χώρες. Αντί 42 TSOs θα έχουμε 5-6 περιφέρειες που θα υπηρετούν, θα εξυπηρετούν τα TSOs. 5 υπηρεσίε θα πρέπει να μοιραστούν. Υπολογισμός δυναμικότητας. Να μην γίνεται κατά χώρα, αλλά κατά περιφέρεια. Και σχεδιασμός για τις διακοπές και τις ελλείψεις, επάρκεια, πρόβλεψη σε περιφερειακό επίπεδο, κοινό, κοινή προσπάθεια και μπορεί να επεκταθεί και το θέλουμε. Όπως σας είπα, αυξάνοντας χρήση ανανεωσίμων χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας. Οι περισσότεροι εθνικοί TSOs αισθάνθηκαν ότι οι καλέ λύσει βρίσκονται σε συνολικό επίπεδο, σε άλλε χώρε, σε γειτονικέ χώρε, μεγαλύτερε περιφέρειες. Αυτό επιδιώκουμε καλή και φθηνή λύση για να εξισορροπήσουμε το δίκτυο. Να έχουμε μια φετηρία, 5-6 περιφέρειες. Προκαθορισμένες υπηρεσίες. Και μπορεί να επεκταθεί. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία, τι στοιχεία μας χρειάζονται, τι δεδομένα χρειαζόμαστε, ρωτήσατε. Ποιο είναι το κόλπο. Θέλουμε να ελευθερώσουμε το δυναμικό του πελάτη, την ευκαμψία διανομής αν θέλετε. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε στοιχεία να ελευθερωθούν, όχι μόνο για τα DSO και τα TSO. Τα DSO και TSO χρειάζονται περισσότερα στοιχεία και θα πρέπει με καλύτερο τρόπο να συλλέγουμε τα στοιχεία προχωρώντας. Οι δεμοί δεν θα ελέγχουμε το σύστημα. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να τρέξουμε το σύστημα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά και υπάρχει μεγάλος πλούτος που υπάρχει που πρέπει να κάνουν κατά υπολογισμούς και επεκτάσεις και προβολές και να αποθηκευτούν τα στοιχεία. Ακούσαμε την παρουσίαση του Βελγίου. Φιλανδία επίσης σύντομα θα έχει κόμβο δεδομένων όπως και ασκανδιναβικές χώρες. Αυτά είναι παραδείγματα συλλογή των στοιχείων για τους πελάτες και έτσι με αυτά μπορούμε να διανύμουμε την ευκαμψία αυτών των στοιχείων, να τρέχει το σύστημα και να αναπτύξουμε και νέες υπηρεσίες πάνω στο σύστημα που παρέχουν την ευκαμψία την απαραίτητη που μπορεί να παρασχεθεί από τα DSOs, TSOs, διεθνώς, εθνικός, όπου υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για την καταβολή του τιμήματος. Τι επίπεδο ευκαμψίας απαιτείται. Η αγορά θα αποφασίσει κατά την απόψή μου. Και είμαστε ένθερμοι υποστηριχτές της αγοράς. Και η ευκαμψία θα προέλθει αποθήκευση από τους πελάτες, από τους διανομείς, από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής, ας αποφασίσει η αγορά. Η ευθύνη για τους TSOs είναι να εξηγήσουν ακριβώς πόση ευκαμψία χρειάζεται στο μέλλον και να αρχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες και μετά θα αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός και οι τιμές και εκείνοι που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες ευκαμψίας θα, πιο φθηνά θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος των αγορών. εκτός μικροφώνου ερώτησης. Ποιος τα αγοράζει? Οι TSOs και τα DSOs τα αγοράζουν την υπηρεσία. Και τα DSOs χρειάζονται την υπηρεσία της ευκαμψίας εξισορρόπησης του δικτύου, αλλά και τα TSOs βέβαια θα αγοράζουν, θα είναι σημαντικοί αγοραστές. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αγορά όπου οι TSOs δεν ελέγχουν, ούτε οι DSOs δεν ελέγχουν. Όλοι μπορούν να βάλουν την υπηρεσία στην αγορά και μπορούμε να ανταγωνιστούμε για να αγοράσουμε τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Εντάξει. Δεν επιτρέπετε, σύντομα να πω κάτι. Στην, η Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια οι πάροχοι παρέχουν την ηλεκτρική ενέργεια, την παρέχουν συνεχώς. Αν δεν μπορούν να παρέχουν αιωλική, θα αγοράσουν από αιωλική. Και ο πάροχος εξισορροπεί τη ροή. Απάντηση. Άλλο μοντέλο έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Έχουμε τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την ισορροπία, που εξασφαλίζουν την ισορροπία. Και αν υπάρχει ανισορροπία, τώρα στην ημερήσια αγορά μπορούν να αγοράσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για να επανεξισορροπήσουν τις θέσεις τους. Αν δεν το κάνουν αυτό θα το κάνουμε εμείς για αυτούς. Και θα τους στείλουμε και τεράστιο τιμολόγιο για αυτή την υπηρεσία. Πολύ ακριβό πολιτική υποστήριξη στην περιοχή. Τι είδους πολιτική στήριξη μπορούμε να φανταστούμε. Αν θέλουμε συντονισμό, την επάρκεια των συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να συνεργαστούν και να συζητήσουν την επάρκεια και η πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο και οι ρυθμιστικές αρχές. Και θα πρέπει να υπάρξει και υποστήριξη, υπάρχει ανταγωνισμός για τα σχήματα υποστήριξης δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος αυτός για να οικοδομήσουμε την πηγή ανανοσίμων ενεργειών. Οι πολιτικοί σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να στηρίξουν την περιφερική υποστήριξη ε, και να είμαστε έτοιμοι με το δίκτυο εν ευθέτω χρόνο και όχι όπως σήμερα όπου έχουμε τις ανανεώσιμες σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιφέρειες που είναι 5-10 χρόνια μπροστά από το δίκτυο, αυτό είναι κάτι κακό που δεν υπάρχει συντονισμό με το δίκτυο. Αναθεώρηση σε ΑΕΣΑ. Τι εντολή μπορούμε να δώσουμε στην Acer. Ανέφερα, αν έχουμε την πρόβλεψη για περιφερειακή επάρκεια και το σχετικό εργαλείο, θα πρέπει να υπάρχει και ρυθμιστικός ρόλος για την Acer να κάνει ελέγχους TSO και DSO να συνεργάζονται για την ε, ευκαμψία της ε, διανομής ίσως χρειάζεται νέα νομοθεσία και αυτό απαιτεί περισσότερη εποπτεία από την Acer Άρα νέοι κανονισμοί, νέες ρυθμίσεις θα χρειαστούν. Τα δίκτυα τα υπεράκτια, offshore networks, θα δούμε τέτοια. Έχουμε πρωτότυπο τέτοιων υπερακτίων δικτύων στην περιοχή μεταξύ Δανίας και Γερμανίας. Θα έχουμε τέσσερις εγκαταστάσεις ολικές και θα συνδέουν τη Γερμανία και την Δανία. Και η Δανία θα αποφασίσει πού θα τοποθετηθούν που θα πουλάει μάλλον ε, την ε, παραγόμενη ενέργεια και θα πουλάει εκεί που είναι πιο καλή τιμή. Είναι ένα πρώτο παράδειγμα. Να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο υπεράκτιο, offshore. Θα επικρατήσει στο μέλλον αυτό. Ναι, μπορεί να μεγαλώσει. Φτιάχνουμε πολλά δίκτυα στη Βόρεια Θάλασσα όπου μπορούμε να κόψουμε ένα καλώδιο αν θέλετε και άμα χρειαστεί να συνδέσουμε μια υπεράκτια ολική εγκατάσταση. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ευελιξία στην Ευρώπη. Θέλουμε να, να έχουμε συστήματα διασύνδεσεως, ε, σημεία επαφής και διασύνδεσης, να μπορούμε να κάνουμε τις προσαρμογές, να κόβουμε κάποια σύνδεση, να βάζουμε άλλη. Τώρα, ροές βρόχου, loop flows, Μπορούμε να, να λύσουμε το πρόβλημα των βρόχων στο μέλλον, ναι. Τι δημιουργεί αυτό το θέμα. Έλλειψη υποδομών και κακοσχεδιασμένες ζώνες ε, δημοπρασιών. Αν έχουμε υποδομές αρκετές στη Γερμανία, δεν θα έχουμε αυτές, αυτούς τους βρόχους που θα δημιουργούνται. Αν έχουμε άλλη δομή για τις ζώνες δημοπρασιών, μπορούμε να το αποφύγουμε για την πρώτη μελέτη των ζωνών δημοπρασιών που θα δημοσιευτεί τον επόμενο χρόνο νομίζω, τον Μάιο-Ιούνιο, θα δείτε ότι θα ξεκινήσει συζήτηση. Θα ανάψει η επιγραφή ε, να δέστε τις ζώνες ασφαλείας όταν δημοσιευτεί αυτή η ε, μελέτη. Από πλευράς TSO πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλες υποδομές για να αποφύγουμε την καταστροφή. Άλλο ένα θέμα. Πρέπει να έχουμε τις σωστές ζώνες τιμολόγησης. Λίγο, λίγο κύριε Πρόεδρε, λίγο ακόμα. Σε προηγούμενο πάνελ απευθύνθηκε έκκληση για μεγαλύτερες ζώνες. Διότι έτσι δημιουργεί το μεγαλύτερο ανταγωνισμό και μεγαλύτερε αλλαγέ. Αυτό είναι αυταπάτη. Διότι η αγορά πάντα σέβεται τους νόμου τη φυσική. Το μόνο θα συμβεί αν έχετε τεχνητή μεγάλη αγορά με εσωτερικές με εσωτερικούς ε, αν θέλετε, ε, τελικά θα γίνεται εμπόριο στο παρασκήνιο και όχι διαφανώς. Όταν θα έχουν κλείσει τα λογιστικά και τα βιβλία θα έχει πολλή δουλειά το TSO. Θα ζητά από τις μονάδες παραγωγής στη Βόρεια Γερμανία να μειώσουν την παραγωγή και από μονάδες στη Νότια Γερμανία να παράξουν περισσότερη ενέργεια. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις τεχνητές ζώνες ε, τιμολόγησης. Υπάρχει λοιπόν μια λύση, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η λύση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω. Όχι στον 22ο αιώνα αυτά όλα, τον 21ο. Ε, ρωτήστε τους αρμοδίους που κάθονται εκεί απέναντι. Με τι με ρωτάτε. Yeah. Ε, κύριος ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω σημειώσει. Ε, σε ό,τι αφορά εμένα, το Data Hub δεν ήταν καμία διένεξη ανάμεσα στους DSO, TSO, τους διαχειριστές δικτύου μεταφοράς ή τους διαχειριστές ε, δικτύου διανομής, ε, ούτε ποιος διαχειρίζεται ποια ε, δεδομένα. Έχει δίκιο ο συνάδελφος ε, θα αυξηθεί περισσότερο η ανταλλαγή των δεδομένων ε, σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στους δύο διαχειριστές έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα των δικτύων μας και ότι θα αντέξουν τα δίκτυα δηλαδή κάθε στιγμή. Με αυτό το Data Hub που δημιουργούμε αν υπάρχει πρόβλημα με τον τελικό διαχειριστή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν έχουμε πέντε data hubs, όπως έχουμε και πέντε clearing houses στο Βέλιο. Ε, έχουμε πέντε διαδραστικές επιφάνειες ε, και ο TSO και όλοι οι προμηθευτές και όλοι οι άλλοι ενεχόμενοι θα πρέπει πέντε φορές να τρέχουν δεξιά και αριστερά για, ε, γι' αυτό τους δημιουργεί περισσότερα λειτουργικά έξοδα. Γι' αυτό εμείς έχουμε ένα σύστημα για όλα τα μέρη, για όλους είναι πιο αποτελεσματικό και για μας και για τον πελάτη ελπίζουμε να είναι διαφανές. Βεβαίως, ε, εάν δεν το αρέσει μπορεί να αλλάξει προμηθευτή. Αλλά ε, τα πέντε clearing houses ε, δούλευαν καλά, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό όταν έχεις ένα data hub και όταν είσαι διαχειριστής δικτύου μεταφοράς. Σημείωσα και μια άλλη ερώτηση για το επίπεδο ευελιξίας. Ίσως να μην είμαι εγώ ο καλύτερος για να απαντήσω ως διαχειριστής δικτύου μεταφοράς. Θα ήθελα να σας πω ότι κάποια στιγμή κάναμε μια μελέτη και ε, κατά ε, για τη μεταφορά στο δίκτυο Βέλγιο ποια είναι η δυνατότητα ε, αποκεντρωμένης ε, παραγωγής στη δική μας περιφέρεια. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι στόχοι που έχουμε στη Φλάνδρα για το 2020 είναι να έχουμε τριπλάσιους πελάτες και πλέον ε, στο βαθμό που λαμβάνουμε υπόψη τον τόπο στον οποίο παράγεται αυτή η αποκεντρωμένη ενέργεια. Τα αποφασίζει η αγορά, το είπε και ο συνάδελφος πώς θα γίνει, αλλά αν πρόκειται για τον τόπο παραγωγής ε, κατά 90-95% μπορεί να είναι όπου θέλει, αλλά και το 5% μπορεί να είναι καλύτερο για την κοινωνία, να είναι μια συγκεκριμένη τοποθεσία μικρή και αποκεντρωμένη. Και αν θέλει ο παραγωγός να σου επιβάλλει τον τόπο παραγωγής, του λέει Εντάξει, αν θες οπωσδήποτε να το κάνεις εκεί και όχι στο 95% που κατά ε, ε, γενική ομολογία αντέχει το δίκτυο, αναλαμβάνει τον κίνδυνο εκείνο. Ε, για να γίνεται όσο είναι περισσότερη ε, παραγωγή με ανανεώσιμες μορφές και που μπορεί κανείς να υποστηρίξει οικονομικά. Και για την ευελιξία, το διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και το διανομέα, υπάρχει μια υπόθεση θα πρέπει να υπάρχει αγορά αυτή. Αν έχουμε πρόβλημα διαχείρισης, συνδιαχείρισης και έχουμε 10 πελάτες μόνο που θέλουν ευελιξία, τότε δεν υπάρχει αγορά. Γνωρίζω ότι σε 10-20 χρόνια μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, μπορεί. Αλλά σήμερα οι δυνατότητες είναι περιορισμένες να το εξάγουμε αυτό ως διαχειριστής δικτύου διανομής. Δεν μιλάω για το μεταφορά τώρα. Ε είναι σχεδόν ανύπαρκτα αυτά σήμερα. Κάποια κυρία ρώτησε προηγουμένως, σήμερα και εμείς εδώ στην περιφέρεια μας δεν έχουμε ε, πάρει απόφαση για τους ε, έξυπνους μετρητές, τα ρολόγια δηλαδή, ε, θα τα ξαναπούμε αυτά. Πολύ σύντομα μπορείτε να μας απαντήσετε ποιος είναι ο βασικός λόγος που, που πριν από λίγο καιρό είχαμε blackout στο Βέλγιο αυτό το ξέρουμε. Ε, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποια πυρηνικά εργοστάσια ε, που ε, έπαθαν βλάβη και αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο, ήταν κάτι απρόπτο, κάτι ξαφνικό και άρχισε ολόκληρη πολιτική συζήτηση για τα πυρηνικά εργοστάσια και ε, υπήρχε και φόβος μήπως έχουμε έλλειψη δεν ήταν blackout αυτό. Ήταν ένα ε, ε, brownout, δηλαδή ήταν ελεγχόμενη η διακοπή ρεύματος αυτό. Ε, δηλαδή, όταν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αυτού του συστήματος του φωτεινού σηματοδότη που κόβει στο ρεύμα επίτηδε σε κάποιες περιοχές για να έχουν άλλες. Ευχαριστώ και πάλι. Δύο ερωτήσεις έγιναν σε μένα η κυρία Κρόβελ για τις επιπλέον αρμοδιότητες που μπορεί κανείς ή θα πρέπει να εκχωρήσει στον Acer, αυτή τη στιγμή όντως ε, ε, με τους κώδικες δικτύων ε, έχουμε νέες οντότητες που δημιουργούνται ή νέα ευρωπαϊκή αγορά με νέους φορείς και διαχειριστές. Αυτοί μπορεί να είναι οργανισμοί που υπάρχουν ήδη και έχουν επιφορτιστεί με το έργο να εφαρμόζουν ε, τους κώδικες των δικτύων ε, σε σημεία που τέμνονται σύνορα κτλ. Ε, όπως είναι το Prismal και άλλες τέτοιες πλατφόρμες που εξορισμού έχουν ευρωπαϊκό ρόλο να διαδραματίσουν και ευρωπαϊκή σημασία. Αυτό θα μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον, γιατί δεν μπορεί ένας φορέας εθνικός ή ένα, ευρω... καθεστώς εθνικό που μπορεί να είναι το γερμανικό, το πολωνικό ή το βελγικό. Οπότε εδώ θα ήταν σκόπιμο ενδεχομένως να το αναλάβει ε, ο Acer. Στο βαθμό που αυτοί οι νέοι οργανισμοί, οι φορείς, πρέπει να ρυθμίζονται από κάπου και κάποιος να τους εποπτεύει. αυτό θα ήταν μια κλασική αρμοδιότητα για τον Acer. Ο ΑΙΣΕΡ δεν είναι μόνο ο οργανισμός που εδρεύει στη Λιουμπλιάνα, είναι και οι εθνικοί ρυθμιστές. Και θα πρέπει κάπως να συμμετέχουν και αυτοί στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Και αν για τη λειτουργία αυτής της πλατφόρμας ή τέτοιων πλατφορμών ε, υπάρχει κάποιο κόστος ε, που επιβαρύνει τους εθνικούς ρυθμιστές, θα πρέπει να αποφασίζουν εκείνοι και να λογοδοτούν και στα δικαστήρια για τις αποφάσεις τους. Και έρχομαι εδώ στην ερώτηση για τη διακυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια συμμετοχή, δηλαδή να μην γίνονται όλα αυτά χωρίς την έγκριση ή χωρίς την πιο έντονη συμμετοχή από ό,τι γίνεται σήμερα του Συμβουλίου Ρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ. Για τις τροπολογίες ε, πρέπει να πω για την έκθεση του κυρίου Λάγκεν έχουμε προθεσμία την 21η Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα. Το απόγευμα, το βράδυ λέει ο κύριος Λάγκεν, απόγευμα. <laughs> Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 7 Απριλίου από 9, 12.30 και 3 με 6.30, 7 ώρες σύνορα και χειροκρότημα παρακαλώ για τους ομιλητές μας. Thank you, thank you very much. For, Ευχαριστώ πολύ θαυμάσια η συζήτηση και οι απαντήσεις καταπληκτικές. Ευχαριστώ όλους τους συνάδελφοι, αγαπητοί βοηθοί, σύμβουλοι και λοιποί παρόντες. Ήταν πραγματικά συναρπαστική η συνεδρίασή μας διήμερη και με